Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στη συνεδρίασή μας. Σας παρακαλώ να καθίστε στις θέσεις σας. Όσοι δεν γνωρίζετε τη γερμανική, να ξέρετε ότι υπάρχει διερμηνία. Τα ελληνικά ακούγονται στην καμπίνα υπαριθμών 7, το νούμερο 7 για τα ελληνικά. Κύριε Λουκά, κύριε Υπουργέ, κύριε Νικολάου. Κύριε Λόπες Αγγουίλιαρ, Πρόεδρε της Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω εδώ σήμερα για τις επόμενες δύο ημέρες του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σας απασχολήσουν ε, θέματα που αποτελούν ίσως ένα από τα πιο δύσκολα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το πακέτο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνήθως θεωρείται ότι είναι ένα βαρετό θέμα, ένα θέμα που απασχολεί μόνο τους ειδικού ή τους ε, πανεπιστημιακούς δασκάλους. Πλην όμως η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους, που μας αφορά όλους. Έχουμε ένα πολύ περίπλοκο πλέγμα καταστάσεων Ε, οι οποίε προκύπτουν ανα πάσα στιγμή θελήσουμε να αγοράσουμε κάτι, να χρησιμοποιήσουμε ένα κινητό τηλέφωνο, να αποστείλουμε δεδομένα από ένα σημείο σε άλλο διότι περνούν ε, τα δεδομένα μα, ε, την χάνουν επεξεργασία μα, από τα κοινωνικά δίκτυα, επί παραδείγματι, από την κοινωνική μα ασφάλιση, από την τράπεζά μα ή από και την, κυβέρνηση μια χώρα. Όταν θέλουμε να κλείσουμε ηλεκτρονικά ένα αεροπορικό εισιτήριο ή οποιοδήποτε άλλο εισιτήριο μεταφορών, τα δεδομένα τα οποία εισάγουμε μπορεί να φτάσουν μέχρι και το σούπερ μάρκετ και να αποθηκευτούν εκεί. Η τεχνολογική εξέλιξη λοιπόν, η τεχνολογική ανάπτυξη, η παγκοσμιοποίηση καθιστούν πολύ πιο ευχερή την συλλογή αλλά και χρήση ως εκ τούτου των δεδομένων. Και άρα έχουν αλλάξει όλο αυτό το πλαίσιο. Νέε λοιπόν μεγάλες προκλήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερω στο πλαίσιο των, ε, της νομοθεσίας του 1995 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να επισημάνω ότι το 1995, από το 1995 πριν από 17 χρόνια μέλος Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ο υποφαινόμενος έλαβε μέρος στην επεξεργασία του εν λόγω νομοθετήματος. Ω μέρο λέει δηλαδή, τη Επιτροπή στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Και πρέπει να σα πω ότι έχω ακόμη στα χέρια μου τα πρακτικά, τα έγγραφα που μα είχαν απασχολήσει σε εκείνη τη συνεδρία του, του 1995. Και ένα πράγμα παραμένει απαράλλακτο, ένα πράγμα παραμένει σταθερό, η ασάφεια, η αδιαφάνεια με το, ε, του νομοθετικού πλέγματος, δηλαδή ο όγκος των δεδομένων που μπορεί κανείς να συλλέξει και να επεξεργαστεί. Αυτό έχει μείνει απαράλλακτο. 12.000 περισσότερα όμως είναι τώρα τα websites. Έχουν 50 κοσταπλασιαστεί ε, οι όγκοι των δεδομένων, 50 φορές δηλαδή περισσότεροι, μεγαλύτεροι είναι οι όγκοι δεδομένων που μεταβιβάζονται, που διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου. Σε ολόκληρη την Ιφίλιο έχουμε κοινωνικά δίκτυα με, 210, με 216 δισεκατομμύρια φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο δίκτυο αυτή τη στιγμή. Είναι αδιανόητο αυτή λοιπόν η τεράστια αλλαγή, η μεγάλη όγκη, η δυνατότητα που θα πρέπει να έχουμε να υπερασπιστούμε, να προασπίσουμε τον προσωπικό μας βίο, καθιστούν πολύ πιο περίπλοκη την κατάσταση, διότι είναι όλο και πιο πολλοί οι χώροι στους οποίους αποθηκεύονται τα προσωπικά μας δεδομένα, στους οποίους εκτίθενται σε πρόσβαση σε τρίτους, ε, στους οποίους την χάνουν επεξεργασίας ανά τον κόσμο και ιδιαίτερως επεξεργασίας είτε πρόκειται για τη διαφημιστική δραστηριότητα, είτε πρόκειται για την εμπορική. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία της προτινόμενης μεταρρύθμισης που απασχολούν φυσικά και εμάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά θα σας απασχολήσουν και εσάς και πιστεύω θα μας στηρίξετε με, την, με τις προτάσεις σας. Ένα πράγμα είναι σαφές βεβαίως, είναι θεμελιώδες δικαίωμα η προστασία των προσωπικών δεδομένων από τον χάρτη των θεμελιωδών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρω ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων που αφορούν στο πρόσωπο του. Άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Η προστασία λοιπόν των προσωπικών δεδομένων δεν είναι μια πολυτέλεια, είναι ένα τμήμα της ταυτότητάς μας και άρα της ατομικής μας ακαιρεότητας, της ακαιρεότητάς μας ως ατόμου μέσα στην Ευρώπη, μέσα στον κόσμο. Είναι ένα χαρακτηριστικότατο ευρωπαϊκό δικαίωμα, ένα δικαίωμα για το οποίο μπορούμε να σεμινόμεθα, ένα δικαίωμα το οποίο ίσως μπορεί να αποτελέσει και πηγή έμπνευση και να εμπλουτίσει ε, τον κατάλογο δικαιωμάτων σε άλλες περιοχές και χώρες του κόσμου. Ένα καινούριο χαρακτηριστικό υπάρχει ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε πλέον αυτό το δικαίωμα και να το προστατέψουμε αποτελεσματικά. Η ουσία, ο πυρήνας του δικαιώματος αυτού είναι η ελεύθερη, ρητή και εξειδικευμένη έγκριση της διαχείρισης των δεδομένων. Αλλά αυτό πώς μπορούμε να το πράξουμε μέσα από το σύστημα, μέσα από το διαδίκτυο, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Πώς μπορούμε επίσης να εξασφαλίσουμε την ε, ουσιαστική προστασία των προσωπικών δεδομένων και των ε, πολιτικών ελευθεριών και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, ε, ειδική αρχή για την προστασία των ατομικών δεδομένων, των, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συγγνώμη, και να τιμήσω το έργο που έχει προσφέρει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προτείνει το συντονισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος με ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση, νομοθετικές πράξεις κατεξουσιοδότηση. Εδώ Θα περιοριστώ σε ολίγες παρατηρήσεις που θεωρώ όμως πολύ σημαντικές. Η απόφαση για την ε, χορήγηση νέων εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τη διαδικασία της των κατεξουσιοδότηση ε, νομοθετημάτων δεν είναι μία κρίση απλή τεχνική, είναι μια πολιτική κρίση η οποία μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την αρχιτεκτονική του συστήματος και γι' αυτό εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη προσοχή θα μεριμνήσουμε, θα επαγρυπνήσουμε ώστε να παρακολουθήσουμε τι περιλαμβάνει η κάθε κατεξουσιοδότηση πράξη και τι δεν περιλαμβάνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ βεβαίως δεν θέλω να το αναφέρω και παρουσία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει από μένα κάθε κατανόηση. Κατανοώ δηλαδή ότι προσπαθεί με ένα ως το δυνατόν μεγαλύτερο όγκο εξουσιοδότηση πράξεων διαφυλάξει τον ρόλο της ως διαχειριστή της νομοθεσίας, ως ε, οργάνου που έχει την πρωτοβουλία της νομοθεσίας, γιατί ε, και αυτό το θεωρώ αυτονόητο πρέπει να σας πω, γιατί κάθε εκτελεστικό όργανο προσπαθεί να διαφυλάξει τις προνομίες και εξουσίες του και στην ε, τοπική μου κοινότητα, όπου ήμουν δήμαρχος, πάλι προσπαθούσε η εκτελεστική αρχή να διαφυλάξει τι ε, αρμοδιότητε και εξουσίε τη. Α, εκ τούτου λοιπόν έχω κάθε κατανόηση για τι προσπάθειε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν αναμένει κανεί από μια εκτελεστική αρχή να εκχωρήσει νομοθετικέ εξουσίε, να παραιτηθεί δηλαδή από νομοθετικέ εξουσίε. Από την άλλη ωστόσο θα πρέπει να μην επαφεθεί μόνη της την κρίση του τι σημαίνει αυτό η κάθε εκτελεστική εξουσία και γι' αυτό ακριβώς έχουμε δικαίωμα να αναπτύξουμε κάθε συζήτηση οπουδήποτε έχουμε να κάνουμε με θεμελιώδη δε δικαιώματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μάτια άργου, με 100 και παραπάνω μάτια θα επαγρυπνεί να εξασφαλίζει ότι έχουμε τη βέλτιστη δυνατή προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, η Επιτροπή από την Επιτροπή των Εσωτερικών των Πολιτικών Ελευθεριών, οι γνωστοί μας, σε όλους μας συνάδελφοι εδώ, είναι μεγάλη ε, προασπιστές των θεμελιωδών ελευθεριών. Σας βεβαιώ ότι την Επιτροπή δεν την βοηθούν καθόλου, την πιέζουν αρκετά, είναι μάλλον άβολοι συνομιλητές. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι καλό να ε, ε, ελέγχεται και το κατά πόσον γνωρίζει ο πολίτης ε, όχι μόνο το να υπάρχουν τα δικαιώματά του, δηλαδή, αλλά κατά πόσο είναι και ο πολίτη ο ίδιο ενήμερο για τα δικαιώματά του. Και σε αυτό ακριβώ εντοπίζεται πρόβλημα και χρειάζεται βελτίωση, γιατί μόνο ένα στου τρει ε, πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι υφίσταται η αρχή προστασία των προσωπικών δεδομένων ή ότι έχει δικαίωμα να ζητήσει την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι εν γνώση του προβλήματος ο πολίτης. Απλώς δεν γνωρίζει ποιες είναι οι υφιστάμενες δομές. 70% του των πολιτών στην Ευρώπη φοβούνται ότι οι επιχειρήσεις συλλέγουν προσωπικά τους δεδομένα και τα χρησιμοποιούν για στόχους διαφορετικούς από αυτούς που αρχικά έχουν ισχυριστεί πως αφορούν. Το ίδιο μεγάλα είναι τα νούμερα και για εκείνου που χρησιμοποιούν τα συστήματα κοινωνική δικτύωσης και εκείνους που κάνουν αγορές μέσω του ίντερνετ. Δηλαδή μεγάλα είναι τα ποσοστά αυτών που θεωρούν ότι δεν έχουν τον έλεγχο επί των προσωπικών δεδομένων. Ε, η δε ψηφιακή γενιά όπως ονομάζεται των 14 έω 25 ετών, οι νέοι αυτοί άνθρωποι, είναι εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά γεννήθηκαν μέσα σε αυτόν τον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης, τον ψηφιακό αυτόν κόσμο, οι οποίοι έχουν πολύ λιγότερη συνείδηση του τι σημαίνουν αυτά τα δικαιώματα ε, από ότι εμείς, εμείς που γεννηθήκαμε στον 20ο αιώνα, στις αρχές, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, έχουν λοιπόν μικρότερη συνείδηση και μικρότερη γνώση των δικαιωμάτων τους. Ταυτόχρονα όμως χρησιμοποιούν πολύ περισσότερα τα μέσα αυτά τα, της κοινωνικής δικτύωσης ή το διαδίκτυο γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ε, τους ενημερώσουμε για τα δικαιώματά τους. Τώρα για την ε, ίδια την πρόταση οδηγίας θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν προτάσεις που αφορούν ε, την ε, κατεργασία προσωπικών, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από ιδιώτες την ε, συλλογή πληροφοριών από τις αρχές ε, της τάξης, την αστυνομία ή τις εγγελικές αρχές, η οποία πλέον είναι πολύ πιο εκτεταμένη από ό,τι πριν από 17 χρόνια, όταν είχαμε την άλλη οδηγία του 1995. Και Φυσικά ξέρουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα συλλογισμών στοιχείων από την αστυνομία τη Αγγελική Αρχή για να μπορούν να επιτελούν το έργο του. Αλλά έχουν και πολύ μεγάλη όρεξη συλλογή δεδομένων, πολύ μεγάλο Πάθο σε αυτή την εργασία συλλογή δεδομένων και γι' αυτό θα πρέπει να το μετριάσουμε. Χρειάζεται δηλαδή μια αναλογική σχέση ως προς τις ε, απαιτήσει για συλλογή δεδομένων που διατυπώνει η αστυνομία ή οι ιδιοκτικές αρχέ γενικότερα. Και επίση θα ήθελα να επισημάνω ότι εγώ ω πρόεδρο του Κοινοβουλίου αλλά και οι δύο συνάδελφοι Δρούτσα και Άλμπρεχτ οι οποίοι είναι εδώ σήμερα συμμερίζονται ξέρω αυτέ τι θέσει ότι ε, τριετία που έχει περάσει από την θέση ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας και την κατάργηση του συστήματος με τους τρεις πυλώνες, έχει φέρει νέα προβλήματα. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν, ε, ότι πολλές φορές το έχω επισημάνει άλλωστε, ότι παραμένουν οι πυλώνες σε ένα βαθμό ε, σε ισχύ, μόνο έξω από, τη, από τις δομές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή δεν μπορεί να τους ελέγξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι πιστεύω ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε μια νέα οδηγία αλλά με τις ίδιες αρχές, με τα, τις ίδιες προδιαγραφές και με την ίδια ισότιμη μεταχείριση των δικαιωμάτων όπως η προηγούμενη του 1995. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι ήδη με τη διαδικασία του Σέγγεν απεδείχθη η αποτυχία της, της ε, κοινοτικής μεθόδου έναντι της διακυβερνητικής. Έγινε προσπάθεια δηλαδή να παραμεριστεί η κοινοτική διάσταση για να ληφθούν οι αποφάσεις διακυβερνητικά. Αυτό απέτυχε το ίδιο πράγμα εάν γίνει προσπάθεια να ε, περάσει με αυτή την οδηγία και πάλι θα αποτύχει. Θα ήθελα να πω δε ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι σημειώνω από την τωρινή προεδρία του Συμβουλίου μεγάλη πρόοδο, αναμένω ακόμη περισσότερες προόδους ε, από την τρέχουσα προεδρία και από την προσεχή προεδρία και εδώ κύριε Υπουργέ θα ήθελα να πω ότι η προεδρία της Κύπρου είναι μια εξαιρετικά καλή προεδρία με πολύ καλή και επικοδομητική συνεργασία μαζί μας. Προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν εντοπίζονται λόγω της τάσης της προεδρίας. Αυτό ήθελα ρητά να το αναφέρω εδώ στη συνεδρίαση. Θέλουμε λοιπόν ένα ενιαίο πρότυπο, θέλουμε ένα Σαφέ ευρωπαϊκό πρότυπο που να ενισχύει τα ατομικά δικαιώματα, που να προαγάγει την εσωτερική αγορά, χωρί ωστόσο να αφήνει δυσανάλογα, χωρίς ωστόσο να επιβαρύνει δυσανάλογα πολύ τι επιχειρήσεις και να μπορεί ταυτόχρονα ο πολίτη και να έχει την πρόσβαση και την εμπιστοσύνη στην πρόσβασή του κατά την ε, χρήση του δικτυακού συστήματο, του ψηφιακού συστήματο, αλλά ταυτόχρονα και να ξέρει ότι, είναι, ε, ότι προστατεύονται τα δικαιώματά του. Στι επόμενε δύο ημέρε, λοιπόν πιστεύω ότι θα μπορέσετε να προχωρήσετε σε μια επικοδομητική και ε, αποτελεσματική ανταλλαγή απόψεων, ε, η μεγάλη πληθώρα ε, παρατηρήσεων, εισφορών, ομιλιών, παρεμβάσεων από τις εθνικές αντιπροσωπείες μας δίνει σαφή εικόνα ότι πρόκειται να γίνει συζήτηση, ότι γενικά έχει αναπτυχθεί ήδη ο δημόσιος διάλογος και, στο, και στα εθνικά αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλετε όλοι να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος μέσω μεταξύ των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορεί να αποτελέσει αυτό υπόδειγμα και για άλλους τομείς ε, νομοθετικούς ότι δηλαδή μπορούμε το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια να εργαστούν συμπληρωματικά μεταξύ τους και με τον Εθνικό Κοινοβουλευτικό Έλεγχο και την Προστασία και με την Ευρωπαϊκή Διάσταση από την άλλη. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε εταίροι τα Εθνικά Κοινοβούλια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή τη νομοθετική. Και έτσι θεωρώ ως εκ τούτου ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διάσκεψή σας. Θα έλεγα σχεδόν ότι ίσως στα 2,5-7 χρόνια της ε, θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η πιο σημαντική διάσκεψη που έχουμε δει. Είναι πολύ σημαντική πάνω απ' όλα διότι έχουμε να κάνουμε εδώ με την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ταυτότητα των κρατών μελών, με την ταυτότητα του πολίτη ως πολίτη της Ένωσης αλλά και ως πολίτη του κάθε κράτους μέλους. Και γι' αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή θα παρακολουθήσουμε τις εργασίες της σκέψεώς σας και γι' αυτό και έρχομαι εγώ ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κηρύξω την έραρξη των εργασιών. Δεν είναι τυχαία η παρουσία μου εδώ. Επέλεξα να είμαι εδώ καθώς ήμουν παλιό μέλος Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών όπως είπα και καθώς αποδίδω ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, έχω ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον στις εργασίες της Επιτροπής αυτής των Πολιτικών Ελευθεριών που είναι στα ε, έμπειρα και ικανά χέρια τώρα του συναδέλφου Λόπε Αγκουίλαρ. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορείτε να και πρέπει να θέστε τα θέματα αυτά των πολιτικών ελευθεριών με πολύ μεγάλη έφαση και ενέργεια και θα ήθελα να ζητήσω κατανόηση από πλευρά σας τώρα για το ότι ίσως χρειαστεί να αποχωρήσω και αυτό δεν θα πρέπει να εκλειφθεί ως έλλειψη σεβασμού και ενδιαφέροντος από πλευρά μου προς το πρόσωπό σας, αλλά ε, να εξηγήσω ότι οφείλεται σε άλλες ελληνικές υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Σούλθ. Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί συνάδελφοι, ευρωβουλευτές και βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων για τις επόμενες δύο μέρες. Αυτή η Διακοινοβουλευτική Επιτροπή θα συζητήσει σε επτά θέσεις. Ξεκινάω με πρακτικές ανακοινώσεις για την οργάνωση. Πρώτα απ' όλα υπάρχει διερμηνία σε 22 επίσημες γλώσσες και τις 22 δηλαδή. Οι εισηγήσει των αγοριτών θα διαρκούν 20 λεπτά συνολικά και μετά θα έχουμε και ερωταπαντήσεις, διάλογο δηλαδή. Θα μπορούν οι βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων και οι ευρωβουλευτέ να θέσουν ερωτήσεις για 45 ή 50 λεπτά κάθε φορά, σε κάθε γύρο συζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παρεμβαίνον θα έχει περίπου πέντε λεπτά ώστε να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του ή να θέσει ερωτήσεις προς τους ομιλητές. Θα μοιραστούν έγγραφα, κάρτες δηλαδή, ώστε να ζητούν το λόγο τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωβουλευτές. Έτσι θα λαμβάνει γνώση ο Πρόεδρος το κατά πόσο θέλουν να θέσουν ερώτηση προς τους παρεμβαίνοντες. Μετά την πρώτη πρωινή μας δηλαδή συζήτηση θα γίνει γεύμα, θα παρατεθεί γεύμα στις 12.30 και το απόγευμα στην απογευματινή συνεδρίαση. Θα συναντηθούμε στις 3 και η εναρκτήρωση εισήγηση θα γίνει από την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ρέντινγκ. Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να σεβαστούν αυτόν τον προγραμματισμό προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχημένα ως τις 7 ε, η συζήτησή μας, καθότι θα παρατεθεί δείπνο στο εστιατόριο των μελών. Όπως σας είπε και ο πρόεδρος Σούλτς, εδώ θα ασχοληθούμε με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό θα είναι και το κύριο θέμα μας, κάτι που απασχολεί τις καθημερινότητέ μα ούτως ή άλλως. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Εδώ οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και παγκοσμιοποίηση έχουν δώσει μια άλλη όθηση στην επεξεργασία των δεδομένων που είναι ευκολότερη και φτηνότερη από ποτεδήποτε στο παρελθόν. Ο όγκος ε, των δεδομένων που συλλέγονται αλλά και η μεταφορά τους ε, και ανταλλαγή τους μεταξύ διαφόρων ε, φορέων και οργανισμών γύρει πολλά ερωτήματα. Αποθηκεύονται, επεξεργάζονται, είναι αντικείμενο επεξεργασία σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει το ε, νέφο ε, ε, του ψηφιακού χώρου ή η αποθήκευση σε μακρινούς, σε, αρχεία στα οποία κανείς δεν έχει εύκολη πρόσβαση και έλεγχο. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν γίνει μέρος της ζωής μας, του καθημερινού μας βίου. Η χρήση επίσης των κοινωνικών δικτύων είναι μια καθημερινή δραστηριότητα. Η επεξεργασία λοιπόν των προσωπικών δεδομένων γίνεται ένα αντικείμενο για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες ακριβώς βάσει της μέρημνας αυτής της επεξεργασίας των δεδομένων. Επίσης επηρεάζονται και οι αρχές ιδιοκτικές επιβολής του νόμου Πολλές φορές αυτό το αναλαμβάνουν και ιδιωτικές εταιρείες. Ε, γύρονται λοιπόν πολλά ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και θα πρέπει να βρεθούν απαντήσεις. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ε, ε, αναφέρεται στην, στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και της ε, στο άρθρο 12 για την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ακριβώς οι προκλήσεις που εμπεριέχει το θέμα. Αυτό είναι και ο τίτλος της διμερίδας μας, η μεταρρύθμιση δηλαδή, του πλαισίου προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων. Το Ευρωκοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σκοπιμότητα των προτάσεων που έχουν τεθεί προς συζήτηση προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων, να εμβαθυνθεί η εσωτερική αγορά, η μείωση του διοικητικού άθους επίσης να επιτευχθεί και να υπάρχει ένας ενίος νόμος που να διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων με συνεπείς μηχανισμούς ελέγχου ε, της νομιμότητας, επιβολής του νόμου δηλαδή. Οι προτάσεις αυτές ενώνονται σε μια δέσμη μέτρων Οπότε υπάρχει πρόταση οδηγίας που ήδη συζητιέται και πρόταση για κανονισμό σχετικά. Και οι δύο εισηγητές ε, βρίσκονται μαζί μας ε, σήμερα και αύριο. Ε, θα παρευρηθούν οι εισηγητές επίσης της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ των πολιτικών ελευθεριών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων μέσα στους επόμενους μήνες θα υποβάλλουν τις δικές τους εκθέσεις. Και μέχρι την άνοιξη του 2013 θα έχουμε μια πρώτη ψηφοφορία ανατολισμού. Τα εθνικά τώρα κοινοβούλια και οι συνεισφορές του θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Είναι καθοριστική σημασία στην όλη νομοθετική διαδικασία. Οι αποκρίσει των εθνικών κοινοβολιών στα ερωτηματολόγια για την προετοιμασία αυτή τη εκδήλωση κιόλα σήμερα υπήρξαν ήδη ιδιαίτερα χρήσιμε. Όλα αυτά εμπλουτίζουν τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και την νομοθετική διαδικασία που διεξαγάγεται εδώ. Και θα πρέπει η τοποθέτησή τους να ληφθεί υπόψη. Η Δημερίδα λοιπόν θα μας δώσει μια συνολική θεώρηση του νομοθετικού, της νομοθετικής δέσμης μέτρων και θα διαφωτίσει και τους συμμετέχοντες. Τώρα, μετά τις ε, ομιλίες των ε, συμμετεχόντων, θα έχουμε, όπως είπα, διάλογο και ευχαριστούμε τους ε, συμμετέχοντες για το ενδιαφέρον και την παρουσία τους. Χωρίς ε, περαιτέρω καθυστερήσεις θα δώσω αμέσως το λόγο στους ε, αγροτές της πρωινής μας συνεδρίασης. Εδώ έχουμε τον Υπουργό Λουκά Λουκά που είναι υπεύθυνο από πλευρά τη Κυπριακή Προεδρία για τα θέματα δικαιοσύνη και δημοσία τάξη. Και έχουμε και τον κύριο Νικολάου μαζί μα, πρόεδρο τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών τη Βουλή των Αντιπροσώπων τη Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουμε επίση εδώ την κυρία Λεμπάγ, Φρανσουά Λεμπάγ, Γενική Διευθύντρια τη Γενική Διεύθυνση ε, Δικαιοσύνη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Ιωνά Νικολάου και θα σας παρακαλέσω να περιοριστείτε σε Mr. President. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, κύριε Λουκά, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Ακουίλα, αγαπητή κυρία Λεμπάιλ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα ενώπιός σας για να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα αυτό της αναθεώρησης του νομικού πλαισίου της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να αναφέρω ότι μόλις πρόσφατα στις 24 Σεπτεμβρίου είχα την τιμή να προεδρεύσω στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων που διεξήχθη στην Κύπρο με θέμα μεταξύ άλλων τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαφύλαξη του δικαιώματος των πολιτών στην ιδιωτικότητα στη ψηφιακή εποχή μέσων σύγχρονων κανόνων για την προστασία δεδομένων η συμπερίληψη του θέματος της αναθεώρησης του νομικού πλαισίου της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στη διάσκεψη αποτελεί ένδειξη της μεγάλης σημασίας που προσδίδει η Βουλή των Αντιπροσώπων στο προτινόμενο πακέτο της Επιτροπής. Στο, στο συνέδριο ανταλλάγησαν ενδιαφέρουσες απόψεις και προβληματισμοί από τους συμμετέχοντες για το προτινόμενο νομικό πλαίσιο. Είναι γεγονός ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από την θέσπιση των υφιστάμενων κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 1993 το διαδίκτυο μετέφερε μόλις το 1% όλων των ηλεκτρονικών πληροφοριών ενώ το 2007 το ποσοστό ήταν περισσότερο από 97%. Η τεράστια εξέλιξη του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια όπως τα υπολογιστικά νέφη, οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσης και οι έξυπνες κάρτες, καθώς επίσης και τα νέα μέσα επικοινωνίας όπως η ισότοπη κοινωνική δικτύωση, η ιστότοπη κοινωνική δικτύωση αποτελούν την καθημερινότητά μας ενώ μας αναγκάζουν να αφήσουμε ψηφιακά ίχνη σε κάθε κίνησή μας. Η διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσων και τις τρίτες χώρες εξελίσσεται ραγδαία. Αν αναλογιστούμε ότι 250 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν σήμερα το διαδίκτυο στην Ευρώπη σε καθημερινή βάση, αμέσως γίνεται αντιληπτό το μέγεθος των προσωπικών μας στοιχείων που φυλάσσονται, διακινούνται και γίνονται αντικείμενων εμπορίας. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και μας καλούν να δράσουμε αποφασιστικά και γρήγορα για να προστατεύσουμε καλύτερα τους πολίτες μας, οικοδομώντας αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην καθημερινή επαφή τους με το διαδίκτυο μόλις το 1 τέταρτο των χρηστών κοινωνικών δικτύων, 26% και ακόμη λιγότεροι αγοραστές μέσω διαδικτύου 18% αισθάνονται ότι έχουν πλήρη έλεγχο των προσωπικών δεδομένων τους. Το 90% των Ευρωπαίων επιθυμεί την αναγνώριση των ίδιων δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. Το 72% των χρηστών του διαδικτύου ανησυχεί για το γεγονός ότι αποκαλύπτει υπερβολικά πολλά προσωπικά δεδομένα και αισθάνεται ότι δεν έχει πλήρη έλεγχο των δεδομένων του. Η φυστάμενη οδηγία χρήζει αναθεώρησης και για τον λόγο ότι η πολυμορφία και ο κατακαιρματισμός που παρατηρήθηκε στην εσωμάτωση και εφαρμογή της από τα 27 κράτη-μέλη έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε νομική αβεβαιότητα με ευρύτερε δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην ενιαία αγορά όσο και στη δημιουργία αναισθήματος εμπιστοσύνης στους πολίτες. Η πρόκληση είναι εδώ. Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο μεταξύ άλλων να κρατά τις ισορροπίες μεταξύ της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ομαλής ρύθμισης της ενιαίας αγοράς. Να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις διαδικτυακές υπηρεσίες να αποτελεί έναν τεχνολογικά ουδέτερο νομικό εργαλείο που να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες αλλά και στις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις, να μειώσει τις γραφειοκρατικές απαιτήσει και το τεράστιο κόστος που αυτή συνεπάγεται, να εξασφαλίσει ομοιόμορφη και ισότιμη εφαρμογή των υποχρεώσεων αλλά και των δικαιωμάτων τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων στα διάφορα κράτη-μέλη. Να μειώσει την διοικητική επιβάρηση που δυσκολεύει την ένταξη πολλών εταιριών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Να καλύψει την διαφαινόμενη αδυναμία της απόφασης πλαίσιων 2008 κάθετος 977, η οποία καλύπτει μόνο τη διασυνοριακή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή λαμβάνοντα υπόψη τις προκλήσεις αυτές, παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2012 πακέτο νομοθετικών προτάσεων το οποίο συζητείται σήμερα την πρόταση κανονισμού που καθορίζει το γενικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων και την πρόταση οδηγίας που καθορίζει κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τη χάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανείχνευσης ή ποινικών αδικημάτων και συναφό δραστηριοτήτων των δικαστικών αρχών. Προτινόμενος κανονισμός επιχειρεί να ενδυναμώσει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών, εισάγοντας νέες έννοιες και ενισχύοντας ήδη υφιστάμενα δικαιώματα. Το δικαίωμα λύθης και το δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή το δικαίωμα σε κάποιον να ζητήσει υπό προϋποθέσεις τη διαγραφή των δεδομένων που τον αφορούν, την απέτηση της ρητής συγκατάθεσης για τη διαχείριση δεδομένων, η διευκόλυνση της πρόσβασης των χρηστών στα δεδομένα τους και η θέσπιση του δικαιώματο φορητότητας δεδομένων δηλαδή η διευκόλυνση της μεταφοράς προσωπικών δεδομένων από έναν πάρχον υπηρεσιών σε άλλον, το δικαίωμα των πολιτών να υποβάλουν παράπονα στην Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων της χώρας τους, ακόμη και όταν ο καθούτο παράπονο εδρεύει σε άλλο κράτος, η καθιέρωση της αρχής της κατασκευής προστασίας της ιδιωτικής ζωής, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνεται υπόψη στο στάδιο σχεδιασμού των διαδικασιών και των συστημάτων. Η εισαγωγή της υποχρέωσης διενέργειας εκτιμήσεων αντικτύπου προστασίας δεδομένων για επιχειρήσεις που διενεργούν επικίνδυνη επεξεργασία. Είναι πρόνοιες σημαντικές και ουσιαστικές προς το επιδιωκόμενο σκοπό. Θα ήταν παράληψη μου να μην κάνω αναφορά στις διατάξεις του κανονισμού που παρέχουν αυξημένη προστασία στους ανήλικους και που προβλέπουν ότι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν παιδιά κάτω των 13 ετών απαιτείται η συγκατάθεση ή η έγκριση του γονέα ή του κηδεμόνα. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών αλλά και των αγορών επιδιώκεται και με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων όπως η εφαρμογή σύγχρονων και ανάλογων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφάλειας, η γνωστοποίηση των παραβιάσεων δεδομένων εντός 24 ωρών από τον εντοπισμό τους, η υιοθέτηση της μονοθυρικής στάσης One Stop Shop, καθιστώντας έτσι υπόλογες της επιχειρήσης σε μία μόνο εθνική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία αυτοί έχουν την έδρα τους όσον αφορά την προτινόμενη οδηγία. Επισημαίνουμε τις ανησυχίες μας που εστιάζονται κατά κύριο λόγο στις διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Ιδιαίτερα τη δημιουργία υποχρέωσης επαναδιαπραγμάτευσης των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες στον τομέα των αστυνομικών και δικαστικών ποινικών υποθέσεων και ειδικότερα όταν αυτές με βάση την εθνική νομοθεσία έχουν κυρωθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι πολυσύνθετο, ευαίσθητο και παράλληλα πολύπλοκο. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και ανησυχίες για το προτινόμενο νομοθετικό πακέτο και γι' αυτό να απαιτείται συνεργασία όλων για να επιτευχθεί η υιοθέτηση ενός νομικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει τις αναγκαίες ισορροπίες μεταξύ της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ομαλής ρύθμισης ενιαίας αγοράς μέσω της ελεύθερης κυκλοφορίας των πληροφοριών. Διακοινοβουλευτικές συζητήσεις, όπως η παρούσα, είναι απαραίτητες και χρήσιμες αφού του ανταλλάσσονται προβληματικοί και σκέψεις για βελτίωση των προτάσεων. Η σημερινή οικονομική κρίση μας σωθεί να εξεύρουμε τρόπον για να εξέλθουμε από αυτήν και μας προσφέρονται το σημερινό νομικό πλαίσιο μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νικολάου, ευχαριστώ πολύ, τηρήσατε πολύ αυστηρά το χρόνο σας, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και τώρα παρακαλώ τον κύριο Λουκά Λουκά, Υπουργό Δικαιοσύνη της ε, ε, Κυπριακής Κυβερνήσεως και Προεδρεύοντα εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο κύριε Λουκά. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής ΛΥΠΕ, κύριε Ακουίλα, αγαπητή κυρία Λεπάη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών του Κυπριακού Κοινοβουλίου, κύριε Νικολάου, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κύριε και κύριοι. Θα ήθελα καταρχά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου για να βρίσκομαι μαζί σα σήμερα σε αυτή τη συνάντηση του Ευρωκοινοβουλίου. Η συνάντηση αυτή καθίστεται ιδιαίτερα σημαντική μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας που αφού μεταξύ άλλων έχει αναβαθμίσει τον ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου ως συνομοθέτη στη διαδικασία υιοθέτηση ευρωπαϊκών νομοθετικών προτάσεων. Το θέμα της σημερινής συνάντησης, δηλαδή προτάσεις της Επιτροπής για την αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποτελεί μια από τις σημαντικές προκλήσεις για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιανουάριο του 2012 η Επιτροπή παρουσίασε το πακέτο προτάσεων για το νέο νομικό πλαίσιο προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιλαμβάνει μια πρόταση γενικού κανονισμού και μια πρόταση οδηγία με σκοπό την ειδική ρύθμιση του θέματο αυτού στον τομέα τη αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει. Οι δύο προτάσει συναταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων τη Κυπριακή Προεδρία λόγω της ιδιαίτερης του σημασία αλλά και λόγω του μεγάλου αριθμού των Ευρωπαίων πολιτών που επηρεάζονται. Η Κυπριακή Προεδρία αντιμετωπίζει τις δύο αυτές προτάσεις ως ένα πακέτο. Είναι γι' αυτό το λόγο που εξετάσαμε και θα εξετάσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων τόσο τον κανονισμό όσο και την οδηγία. Να υπενθυμίσω ότι η πρόταση κανονισμού καταργεί την οδηγία 46 του 1995 που αποτελεί το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τροποποιεί την οδηγία του 2002, 58 του 2002 που προνοεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η θέσπιση του νέου νομικού πλαισίου κρίθηκε απαραίτητη λόγω της ανάγκης καλύτερης αντιμετώπισης των προκλήσεων που παρουσιάζουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση αλλά και λόγω της υποχρέωσης εναρμόνισης με τις νέες υποχρεώσεις που επιβάλλει η συνθήκη της Λισαβόνας. Με την πρόταση αυτή, η Επιτροπή επιδιώκει να διασφαλίσει ένα ψηλότερο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενδυναμώνοντας τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα των ανήλικων χρηστών του διαδικτύου. Επιπρόσθετα, αποσκοπεί στο να επενδύσει στην εμπιστοσύνη του ώστε να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικός παίχτης στη, στη σημερινή ψηφιακή οικονομία και να εδραιώσει τη θέση τη στο διεθνή χώρο τη διασυνοριακής ροής των πληροφοριών. Ως Προεδρία, εργαζόμαστε στην επίδεξη, προς αυτού του στόχου. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες, όλες τις ανησυχίες, κρατώντας τις ισορροπίες προς κάθε κατεύθυνση. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το νέο νομικό πλαίσιο αναμένεται ότι θα ρυθμίζει τα επόμενα χρόνια την προσωπική μας ζωή, την αγορά, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις. Γι' αυτόν τον λόγο η Προεδρία στοχεύει στο να παραδώσει στη μελλοντική Προεδρία, την Ιρλανδία, ένα ποιοτικό έργο στη βάση του οποίου θα μπορεί να συνεχίσει και αυτή με τη σειρά της της προσπάθειας. Όπως γνωρίζετε, ο κανονισμός εφαρμόζεται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Εισάγει καινοτόμε έννοιε όπω το δικαίωμα λήθης, δηλαδή το δικαίωμα κάποιου, για παράδειγμα, να ζητήσει τη διαγραφή μια φωτογραφία του από το διαδίκτυο και την περαιτέρω επανεδημοσίευση τη σε άλλε ιστοσελίδε. Εισάγεται επίση η αρχή τη λογοδοσία, δηλαδή η υποχρέωση κάποιου υπεύθυνου επεξεργασία να συμμορφώνεται αλλά και να επιδεικνύει τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του κανονισμού. Μια άλλη σημαντική αναβάθμιση που εισάγει, ο κανονισμός είναι ο όρος της μονοθυρικής στάσης, one-stop shop, που στοχεύει στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, καθορίζοντας ότι κάθε πολίτης θα απευθύνεται μόνο σε μια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων ενώ ταυτόχρονα και οι επιχειρήσεις θα είναι υπόλογες σε μια μόνο αρχή. Περαιτέρω προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού συνοχής, με τον οποίο θα διασφαλιστεί η δυνατότητα ανάληψης κοινών δράσεων των εποπτικών αρχών, η ομοιόμορφη επιβολή κυρώσεων και η επίλυση διαφορών όπου προκύπτουν. Επιπρόσθετα, ο κανονισμό δημιουργεί στου κατασκευαστέ και στου υπεύθυνου επεξεργασία καινούριε υποχρεώσει για προστασία τη ιδιωτικότητα όπω το privacy by design, δηλαδή την εισαγωγή μέτρων προστασία στο στάδιο σχεδιασμού μια καινούρια τεχνολογία και την υποχρέωση πραγματοποίηση ειδική έκθεση αντιχτύπου privacy impact assessment πριν την εφαρμογή των μέτρων που συνεπάγονται κάποια παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή. Οι μέχρι τώρα συζητήσει τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο έχουν καταδείξει ότι το κείμενο του κανονισμού χρειάζεται βελτίωση και προ αυτήν την κατεύθυνση, ε, εργαζόμαστε. Είναι παραδειχτό από όλου μα ότι χρειάζομαστε ένα ξεκάθαρο κείμενο, ένα ξεκάθαρο νομικό εργαλείο χωρί ασάφειε και γκρίζε ζώνε. Πρέπει να αποφύγουμε καταστάσει οι οποίε στο μέλλον μπορεί να οδηγήσουν σε αδιέξοδα επιφέροντας πλήγμα στην τεχνολογική ανάπτυξη, στην ίδια την αγορά, στη βιομηχανία, αλλά και στους ίδιους τους πολίτες μας. Τώρα όσον αφορά την πρόταση οδηγίας, όπως γνωρίζετε καλύπτει την επεξεργασία και ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων που γίνεται από τις αρχές επιβολής του νόμου σε εθνικό επίπεδο, σε διασυνοριακό επίπεδο μεταξύ των αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες. Η οδηγία θα αντικαταστήσει την απόφαση πλαίσιο του 2008-977, η οποία σήμερα καλύπτει μόνο την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρχών κρατών μελών και τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες. Από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εξαιρούνται τα όργανα της ε, Ένωσης, όπως η Europol και η Eurojust και οι μυστικές υπηρεσίες. Η αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου κρίθηκε αναγκαία λόγω των υποχρέωσεων που απορρέουν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα, που επιβάλλουν όπω οι κανόνε προστασία προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται σε όλου του τομεί τη Ένωση, περιλαμβανομένου και του τομέα τη αστυνομική και δικαστική συνεργασία, σε ποινικέ υποθέσει και λόγω τη ανάγκη ενδυνάμωση τη συνεργασία και τη επιχειρησιακή ικανότητα των αρχών επιβολή του νόμου. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, η οδηγία έχει, εξετάσει, έχει εξεταστεί σε τεχνικό επίπεδο τον Σεπτέμβριο και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί κατά τους επόμενους μήνες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν για την οδηγία, όμως οι προσπάθειες σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν. Επίσης είναι γνωστές οι επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί στο Συμβούλιο αλλά και ο προβληματισμός που επικρατεί γενικότερα Παρ' όλα αυτά, στηρίζουμε τι εργασίε μα για την οδηγία και σε στενή συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Συνεχίζοντα, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι σε τεχνοκρατικό επίπεδο οι εν λόγω προτάσει συζητούνται στην ομάδα εργασία TEPIX του Συμβουλίου. Η Κυπριακή Προεδρία προγραμμάτισε έξι διμερεί συναντήσει για τι συζητήσει του. Παράλληλα, ορισμένα οριζόντια θέματα που προέκυψαν κατά τη συζήτηση τη πρόταση κανονισμού και διαφάνηκε ότι απασχολούσαν όλα τα κράτη-μέλη, παραπέμφθηκα για συζήτηση στο άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στη Λευκοσία. Για πολιτικό προσανατολισμό, τον περασμένο Ιούλιο στη Λευκοσία. Το Συμβούλιο ΔΙΕ εξέδωσε ξεκάθαρη εντολή για διερεύνησή του και το λόγο αυτό η Κυπριακή Προεδρία προγραμμάτισε αριθμό συναντήσεων των φίλων της Προεδρίας. Για να συντομεύσω την ομιλία μου, κύριε Πρόεδρε, να αναφέρω ότι τα θέματα αυτά που απασχόλησε το Συμβούλιο ήταν το διοικητικό κόστο όσον αφορά τι μεσαίε και μικρέ επιχειρήσει, τι διατάξει του κανονισμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και, μεγάλο αριθμό, και ο μεγάλο αριθμό ε, πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Όπω έχει αναφέρει και ο πρόεδρο Σούλτ, όλα τα κράτη-μέλη απασχολούν αυτό το θέμα. Κλείνοντα, θα ήθελα να τονίσω ότι για επίδεξη των στόχων μας η συνεργασία μαζί σας είναι απαραίτητη και αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της επιτυχίας μας. Θεωρούμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι ο βασικός εταίρος μας. Έτσι θα πρέπει να εργαστούμε μαζί και συλλογικά για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε σήμερα ένα νομικό εργαλείο όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα το οποίο να, να ενισχύσει τις αρχές που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ταυτόχρονα να αποτελεί το εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Luca. Now the third floor goes to François Ευχαριστούμε κύριε Λουκά και τώρα λόγω στην κυρία Λεμπαΐλια, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης. Well, thank you. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θέλω να πω ότι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλωσορίζουμε τον διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Βεβαίως, γνωρίζουμε ότι συνεισφορές έχουν ήδη υποβληθεί από αρκετά από αυτά τα κοινοβούλια και θα λάβουμε σοβαρός υπόψη τις προτάσεις, τα σχόλια που έχετε ήδη κάνει. Η διάσκεψη αυτή νομίζω οργανώθηκε την κατάλληλη χρονική στιγμή. Διότι έχουμε ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με τον σύνομοθέτη μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οπότε με τις συνεισφορές σας σήμερα θα εμπλουτίσετε σημαντικά τον διάλογό μας. Ακούσατε ήδη από το πρωί πολλά για την προστασία των δεδομένων. Αυτό που θα ήθελα να κάνω από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προσπαθήσω να ανακεφαλαιώσω το τι προθέσεις είχαμε όταν υποβάλαμε τις προτάσεις μας και για την οδηγία και για τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Νομίζω μέρος της απάντησης εμπεριέχεται στον τίτλο ακριβώς της διάσκεψής μας ή μάλλον της πρωινής Συζήτηση. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνη σε έναν ψηφιακό κόσμο. Μια παγκοσμιοποιημένη υφήλιο. Ακούσατε τους ε, αγορητέ μα να λένε πόσο η επεξεργασία δεδομένων εξελίσσεται και πρόκειται να εξελιχθεί περαιτέρω τα ερχόμενα χρόνια. Πρώτος λοιπόν ε, στόχος που είχαμε υπόψη μας κατά την επεξεργασία της πρότασής μας ήταν να ενδυναμώσουμε τα ατομικά δικαιώματα. Θέλουμε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν τα δεδομένα τους. Γι' αυτό ακριβώς προτείναμε το δικαίωμα στη λύθη, όπως ονομάστηκε, τη φορητότητα των δεδομένων, την, το δικαίωμα σε αντίτυπο των δεδομένων και τη μεταφορά τους σε άλλων παροχέα υπηρεσιών. Προτείναμε επίσης μέτρα διαφάνειας ε, σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή, ένας πολίτης, ένα άτομο να μπορεί να γνωρίζει μια εταιρεία, ένας δημόσιος φορέας, τι διαθέτει από τα προσωπικά του δεδομένα στα χέρια της ή στα χέρια του. Νομίζουμε λοιπόν αυτοί οι όροι μπορούν ακριβώ να μα επιτρέψουν να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη σε ένα ψηφιακό κόσμο. Οι λόγοι για όλα αυτά είναι για να προστατε... που γίνονται όλα αυτά είναι για να προστατεύσουμε ακριβώ του πολίτε. Θεωρούμε ότι είναι ακόμη και ζήτημα εμπορική σημασία το να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη στον ε, ψηφιακό κόσμο. Οι επαφέ, οι συνομιλίε που είχαμε από τότε που αρχίσαμε να μελετούμε την πρόταση αυτή, ακριβώ αυτό μα δείχνουν. Ότι ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών δηλαδή, επειδή ακριβώς δεν εμπιστεύεται τον ψηφιακό κόσμο, το ψηφιακό περιβάλλον, επιφυλάσσεται, δεν κάνει αγορές στο διαδίκτυο ή δεν επιτρέπει την ε, αποστολή δεδομένων του για διάφορους σκοπούς. Αυτός λοιπόν ήταν ο πρώτος στόχος που είχαμε κατά νου, η προστασία των πολιτών, των ατομικών δικαιωμάτων, καθώς και η οικοδόμηση εμπιστοσύνη ένα ψηφιακό περιβάλλον. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν να απλουστεύσουμε το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων. Εάν ρίξετε μια ματιά στο τι συμβαίνει στον χώρο τη προστασία των δεδομένων, αυτό το διάστημα θα δείτε ότι υπάρχουν 27 διαφορετικά καθεστώτα ε, συστήματα προστασία των δεδομένων. Ακριβώ διότι δεν υπάρχει υπάρχει μάλλον μόνο μια οδηγία που ισχύει, η οποία ήταν ένα ορόσημο στην εποχή τη κατά την ε, εξέλιξη των αναγκών προστασία των δεδομένων, όμω η οδηγία αυτή έχει μεταφερθεί με διαφορετικού τρόπου, όπω συνήθω συμβαίνει με τι οδηγίε με διαφορετικούς τρόπους στα 27 κράτη-μέλη. Αυτό δυσκολεύει τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Εάν είναι κανείς εταιρεία ή επιχείρηση που εργάζεται σε αυτό το χώρο, έχει ανάγκη να γνωρίζει το τι ισχύει στην νομοθεσία του κάθε κάτω μέλου και πρέπει να ασχολείται και με τι ε, απαιτήσει των αρχών προστασία των δεδομένων. Όλα αυτά πρέπει να ευθυγραμμιστούν λοιπόν. Ο τρόπο που σκεφτήκαμε να το κάνουμε αυτό είναι η επιλογή του εργαλείου. Επιλέξαμε λοιπόν τον κανονισμό, ο οποίο ε, εφαρμόζεται άμεσα και σκεφτήκαμε να υπάρχει ένα νόμο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι θα επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν ε, τουλάχιστον ένα δις ευρώ ετησίως με την ύπαρξη ε, μία ενιαία νομοθεσία. Η δεύτερη πτυχή που συνοδεύει και προστατεύει του πολίτε είναι να υπάρχει μια κοινή αρχή προστασία των δεδομένων. Έτσι, οι επιχειρήσει και οι εταιρείε που λειτουργούν σε διαφορετικά κράτη-μέλη θα ωφεληθούν ε, τα μέγιστα. Διότι θα απευθύνονται σε μία και μόνη ε, αρχή προστασία των δεδομένων στον τόπο της κύριας εγκατάστασης. Αυτά για τους ε, σκοπούς απλούστευσης. Κάτι άλλο που είχαμε κατά νου επίσης ήταν να βεβαιωθούμε ότι όταν θα θεσπίσουμε τα διοικητικά μέτρα που χρειάζονται για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το όλο σύστημα, θα φροντίσουμε να υπάρξει και ιδιαίτερη μεταχείριση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι το 99% των εταιριών μας είναι τέτοιες. Και ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν βεβαίως, αλλά θέλουμε να μειώσουμε για αυτές το διοικητικό άχθος. Θα δείτε στις προτάσεις μας ότι υπάρχουν πολύ στοχευμένα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υποχρεώνται να έχουν υπάλληλο προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων ή να διεξαγάγουν μελέτε αντικτύπου ή να ετοιμάζουν ε, την τεκμηρίωση που απαιτείται από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Βέβαια υπάρχει μια εξαίρεση εδώ. οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ακριβώς ασχολούνται με την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Όμως τεράστια πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απελευθερώνονται ακριβώς από το βάρος αυτό. Από το άχθος αυτών των απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Ο επόμενος στόχος που είχαμε κατά νου ήταν να έχουμε μια ασφαλή νομοθεσία. Εάν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα εγκρίνουμε νομοθετικό πλαίσιο, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να αντέξει και στο χρόνο, να είναι ασφαλής για το μέλλον. Να μην χρειάζεται να γίνει αναθεώρηση σε μια διετία. Να λέμε σε δύο χρόνια οι ανάγκες μας ξεπέρασαν, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και να γίνονται συνεχεί μετατροπέ. Όχι. Θέλουμε ε, μια νομοθεσία που να διαρκέσει. Γι' αυτό ακριβώς προτείναμε μια σειρά από μέτρα. Μέτρα που θα μας επιτρέψουν να το πετύχουμε αυτό. Ένα από αυτά αναφέρθηκε και από τον πρόεδρο Σούλτ το πρωί. Η κατεξουσιοδότηση πράξη. Να πω δύο λόγια για αυτό το θέμα. Αυτές οι πράξεις μας δίνουν τη δυνατότητα σε εμά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνουν τη δυνατότητα βάση του κανονισμού και υπό την επαγρύπνηση βεβαίω του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου να εξηγήσουμε λεπτομέρειες, να διευκρινίσουμε στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό. Δεν αναθεωρείται έτσι όμως ο κανονισμός, διευκρινίζεται. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε τις εξουσιοδότηση πράξεις ως ένα μέσο που μας επιτρέπει να είμαστε ευέλικτοι, εάν θέλουμε νομοθεσία που να αντέξει στο χρόνο. Υπάρχουν λοιπόν σχετικές διατάξεις, αλλά καθώς δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να κάνω δύο σχόλια και για την οδηγία. Η οδηγία επικεντρώνεται στην επιβολή του νόμου, στην φορητότητα, τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα. Και νομίζουμε ότι σε σχέση με την απόφαση πλαίσιο που ήδη ισχύει, η πρόταση που έχουμε θέσει επιτάπητος αποτελεί μια πραγματική βελτίωση. Ο τρόπος υλοποίησης υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ήδη ένα τέτοιο βήμα, κάτι που δεν ισχύει για την υπάρχουσα νομοθεσία. Επίσης, η οδηγία κατά τη διαστολή ως προς την απόφαση πλαίσιο καλύπτει όχι μόνο τα διασυνοριακά ζητήματα, αλλά και την ε, ε, εσωτερική, την εγχώρια επεξεργασία δεδομένων από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Ο κύριος λόγος ήταν ότι είναι όλο ένα και πιο δύσκολο να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του διασυνοριακού και του εγχώριου στοιχείου. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι με τους οποίους το συζητήσαμε το θέμα αυτό ε, λένε ότι είναι σχεδόν ανέφικτο. Επιλέξαμε λοιπόν να καλύψουμε και τις δύο αυτές διαστάσεις τη διασυνοριακή και την εσωτερική. Επίσης, επιδιώκουμε να εναρμονίσουμε τους περιορισμούς τους γενικούς κανόνες. Προς στιγμή, οι περιορισμοί στους γενικούς κανόνες είναι δικαιολογημένοι, ιδίως στον τομέα της επιβολής. Και είναι βεβαίως διαφορετική από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Αυτό που ακριβώς προτείνουμε είναι να υπάρξει εναρμόνιση αυτών των κριτηρίων των κριτηρίων ε, για τις εξαιρεσει και για τον περιορισμό των ε, δικαιωμάτων των πολιτών. Ακριβώς με τις διατάξεις αυτές θέλουμε να εφαρμοστεί η αρχή της προστασίας των δεδομένων και στον τομέα επιβολής του νόμου, δηλαδή εκεί που βρουν οι αρχές. Βεβαίω με όλο τον απαραίτητο βαθμό πρόληψη, γιατί είναι ένα ευαίσθητο τομέα. Ε, επιτρέψτε μου να συμπεράνω ότι η συνεργασία μας με τους συνομοθέτες μας είναι ιδιαίτερα επικοδομητική. Και όπως είπαν και οι υπόλοιποι ομιλητές μας, πραγματικά υπάρχει στήριξη προς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες αμφιβολίες, απορίες, εγείρονται κάποια ζητήματα. Αυτά όμως με τρόπο ιδιαίτερα επικοδομητικό θα φροντίσουμε να τα επιλύσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Αλεμπάη. Και τώρα ακούμε παρεμβάσεις. Πέντε συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. Θα ξεκινήσουμε, θα τους ακούσουμε όλους και μετά θα γυρίσει ένας τελικός γύρος ε, απαντήσεων ίσως από τους ε, παρισταμένους εδώ στην έδρα. Η κυρία Μπαντέτ από την Βουλή, την, από ε, την Γερουσία της Ισπανίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και συγχαρητήρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει οργανώσει αυτή τη ε, συνεδρίαση και δίνει τη δυνατότητα σε εμά από τα Εθνικά Κοινοβούλια να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος και να συμβάλλουμε σε αυτό το διάλογο. Να κατα... Καταρχήν να συγχαρώ την Επιτροπή για την πρωτοβουλία της αυτή, νομοθετικής φύσεως, για αυτό το θέμα της αναθεώρησης των ε, ε κανόνων του νομοθετικού πλουσίου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των δεδομένων. Σε γενικέ γραμμέ είναι θετικό βλέποντα τον όγκο των πληροφοριών που έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Έχουμε τα κριτήρια τα εδαφικά και αυτά έχουν ξεπεραστεί θα λέγαμε. Όλα λειτουργούν διαδικτυακά. Επίση είναι θετικό για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο συντονισμένη ε, προσέγγιση από τις χώρες μέλη. Η οδηγία του 95 έχει μεταφερθεί, ενταχθεί στα επιμέρους ε, νομικά πλαίσια των χωρών, όχι με ομοιόμορφο τρόπο. Επίσης, να πω ότι μας είναι θετική αυτή η προσέγγιση, διότι συγκεκριμενοποιεί το πλαίσιο, το κανονιστικό και ξεπερνάει κανείς το αόρια, τα αυστηρά όρια της ε, ευρωπαϊκής επικράτειας. Τώρα, υπάρχουν δύο στόχοι σημαντικοί τώρα. Ξάλλου έχουν, τα έχουν αναφέρει. Απ' τη μια, θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικότητα, να υπάρχει ουσιαστική προστασία των πολιτών και να δίνει την κατάλληλη ασφάλεια στις επιχειρήσεις. Επιπλέον αυτό το όργανο θα πρέπει να έχει διάρκεια. Γι' αυτό η νομοθεσία δεν θα πρέπει ε, να περιορίζεται στις τεχνολογικές ε, εξελίξεις και σε αυτά τα μέσα διότι έξι θα ξεπεραστεί αργά ή γρήγορα. Ο κύριος Νικολέα αναφέρθηκε στο θεμα της ε, ε Η νομοθεσία θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και θα πρέπει να την ξαναδούμε, να την ξανααναθεωρούμε. Στον κανονισμό Φελπίν, το άρθρο 17 ε, για το δικαίωμα της λύθης Έχουμε άλλη διαφορετική ολογία σε ισπανικά για αυτή την έννοια. Θα ήθελα να ξέρω την άποψη των μελών εδώ στο βήμα σε σχέση με την υψίουσα νομοθεσία. Διότι υπάρχει θέματα, υπάρχουν θέματα ευθύνη χωρίς να προσδιορίζονται αυτά. Ε, οι ερευνητές, ό,τι χρησιμοποιείται σε όλα αυτά, τη διαδικασία δεν είναι ουδέτερη. Θα πρέπει να δώσουμε μια έμφαση βασικά όλα να συγκλίνουν προς την προστασία του πολίτη. Διότι τα πράγματα μπορούν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου δεν έχουμε την κατάλληλη προστασία του πολίτη. Στα πλαίσια τώρα της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης που έχουμε, είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την δημοκρατική και διαθεσμική διάσταση. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε όλες αυτές οι πράξεις προβλέπονται ε, θα πρέπει να γίνει κατανοητό δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα με πράξεις οι οποίες έχουν καθαρά νομοθετικού χαρακτήρα οι οποίες εφαρμόζονται. Θα πρέπει δηλαδή να προβλεφθούν πράξεις οι οποίες να έχουν καθαρά μια δημοκρατική διάσταση. Ευχαριστώ. Mm. Ευχαριστούμε κυρία Αλεγκρίνη. Ευχαριστώ. Η Ιταλία είναι σίγουρα υπέρ του καθεστώτος προστασία των προσωπικών δεδομένων, με κάποιε βεβαίω επιφυλάξει. Θεωρούμε ότι υπάρχουν και κάποια όρια. Ε, στα εργαλεία που θα πρέπει να προβλεφθούν, στα μέτρα που θα διέπουν τον ποινικό τομέα για τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, δηλαδή τις διατάξεις που θα αφορούν τη Europol και τη Eurojust. Βεβαίως η, θετική, η αποτίμησή μας γενικώ είναι θετική. Θα πρέπει να ορίσουμε υψηλότερε προδιαγραφές που να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την ε, επικράτεια ομοιόμορφα αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα και την αρχή τη επικουρικότητας και τα κριτήρια που αυτή επιβάλλει. Θα πρέπει να υπάρξουν και συνταγματικές μεταρρυθμίσεις σε κάθε χώρα ή σε πολλές περιπτώσεις για να μπορέσουν να ισχύσουν όλα τα μέτρα που προβλέπονται. Έπειτα, ο ορισμός ομοιογενών προτύπων μπορεί να ε, υποβαθμίσει το επίπεδο προστασίας κάποιων ε, εθνικών συστημάτων που είναι ήδη εξελιγμένα. Να περιοριστούν δηλαδή τα υπάρχοντα εχέγγυα σε ορισμένες χώρες. Επίσης, η πρόταση αντιφάσκει με την αρχή της επικουρικότητας λόγω και των όσων προβλέπει το άρθρο 87 με τις ε, εκορίσεις αρμοδιοτήτων. και τη μεταφορά δεδομένων λόγου χάρη σε τρίτε χώρε που είναι κάτι το ιδιαίτερα επικίνδυνο. Πάλι στο άρθρο 51 υπάρχει αντίφαση με την αρχή της επικοτικότητα, όπου γίνεται λόγος για τη μοναπευθυντική θηρίδα. Εκεί οι πολιτε μπορούν να απευθυνθούν στην αρχή ελέγχου της ε, κάθε χώρας. Μια άλλη αντίφαση προκύπτει από το γεγονός ότι εφόσον ο κανονισμό υποκαταστήσει την ισχύουσα οδηγία και η ισχύ του θα είναι ευρύτερη από τη οδηγία, θα πρέπει ακριβώ να είναι και πιο συγκεκριμένο. Όπω στην περίπτωση του άρθρου 17 το δικαίωμα στηλήθηκε, στο άρθρο 21 την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, διότι εκεί θα μπορούσαν να προκύψουν διαφορές ή κλίμα νομικής αβεβαιότητας στα κάτι μελη Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Και τώρα από το Πολωνικό Κοινοβούλιο ο κύριος Κάλιστ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και επιτρέψτε μου να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία της και να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για την συνεδρίαση σήμερα. Εμείς στην Πολωνία είμαστε υπέρ των προτάσεων καθώς πρέπει να εξασφαλιστεί ένα αποτελεσματικό και σύγχρονο σύστημα δίκτυο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αλλά όπου υπάρχουν ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις πρέπει οπωσδήποτε να ερμηνεύσουμε ώστε αυτές να έχουν ρητά προβλεφθεί. Να μην υπάρχει υπερβολική δηλαδή ανάθεση στη διαδικασία των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων, γιατί αυτό σημαίνει ότι ε, παραγωνίζουμε τα κοινοβούλια. Το άρθρο 17 ιδιαίτερος θα ήθελα να υπογραμμίσω λοιπόν το δικαίωμα του να λησμονηθεί κανείς, το δικαίωμα στη λύθη δεν προβλέπεται που ρητά. Δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Και στην εποχή την ψηφιακή, στην εποχή του ίντερνετ, του διαδικτύου, εκεί όπου, εδώ μάλλον, που μέσα σε δευτερόλεπτα εμφανίζονται ε, ιστοσελίδες, η αναφορά σε ένα τρίτο μέρος είναι υπερβολικά ασαφής, δεν προσφέρει επαρκή προστασία. Επίσης υπάρχει μια παραπομπή στο άρθρο 2, ωστόσο η συνθήκη χωρίζεται σε κεφάλαια και από εκεί και κάτω σε, σε τίτλους και μετά σε κεφάλαια. Ε, έτσι λοιπόν δεν είναι καθόλου σαφές όταν γίνεται παραπομπή στο κεφάλαιο 2, σε ποιο κεφάλαιο, ποιανού τίτλου αναφέρεται. Βλέπω ότι είναι κακογραμμένο το κείμενο. Επίσης η δυνατότητα διαχείρισης μάλλον προστασία σε πρώτος διαχείρισης από διαχειριστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα επιληθεί. Το θέμα της γλώσσας επίσης. Εφαρμόζεται αυτή η αρχή προσωρινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Εμείς στην Πολωνία έχουμε κάποιες δυσκολίες σχέσεις με τις διεθνείς συνθήκες, καθώς κάποιοι εκ των γειτόνων μας, Φερρυπίν Ρωσία, αξιοποιούν προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εξυπηρετήσουν το ολοκληρωτικό τους καθεστώς. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε υπόψη. Και γι' αυτό νομίζω θέλει πολύ ακόμη δουλειά αυτό το σχέδιο. Ο κύριος Τριανταφυλλίδη, παρακαλώ εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακόμα δύο λεπτά. Θέλω να καλωσορίσω τους δύο διακεκριμένους ε, ομιλητές, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον ε, κύριο Νικολάου της Κυπριακής Βουλής. Ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, αν λάβουμε υπόψη την, ε, τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Νικολάου, φαίνεται ότι η αναθεώρηση του πλαισίου είναι όσο πιο επίκαιρη μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, Όλοι σήμερα χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, όλοι χρησιμοποιούμε τα έξυπνα τηλέφωνα, τις ταμπλέτες, το online banking κλπ. Η παρατήρηση μου είναι ότι ε, παρόλο που είναι τόσο επίκαιρη η αναθεώρηση, μου φαίνεται πως προχωρεί υπερβολικά αργά. Το δεύτερο μου σχόλιο είναι ότι θα αναμέναμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ισχύσει ένας γενικός κανονισμός ο οποίος να θέτει ένα σαφές νομικό πλαίσιο και αντί αυτού καταλήγουμε να έχουμε έναν κανονισμό και μια οδηγία. Αυτός ο κατακαιρματισμός μου φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα περιθώριο για ελιγμούς και παραθυράκια, ενώ αυτά ακριβώς είναι που προσπαθούμε να αποφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η τάση προς τη δημιουργία εξαιρέσεων μπορεί επίσης να παρατηρηθεί στο ίδιο το περιεχόμενο του πακέτου για την προστασία δεδομένων μέσω τη χρήση γενικών ορισμών όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται για την ταυτότητα του προσώπου, το έννομο συμφέρον ή και το δημόσιο συμφέρον. Αλλά πώς μπορούμε να μιλάμε περί δημιουργίας εμπιστοσύνης σε ένα ψηφιακό κόσμο, εάν οι κανόνες του παιχνιδιού είναι ασαφείς λόγω εξαιρέσεων. Και το τρίτο σχολείο, ακόμη και αν γινόντουσαν δεκτά αυτά τα διαφορετικά εργαλεία, οι σημαντικά χαμηλότερες προδιαγραφές της οδηγίας που αφορά τις αρμόδιες αρχές για ποινικά αδικήματα είναι προβληματικές. Ιδιαίτερα σήμερα όπου οι αρχές επιβολής του νόμου αναζητούν όλο και περισσότερη πρόσβαση στις βάσεις προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από ιδιωτικούς φορείς. Και τέλος κύριε Πρόεδρε ήθελα να ρωτήσω πώς δικαιολογεί το Συμβούλιο αυτών των κατακαιρματισμών και δεύτερον πότε μπορούμε να περιμένουμε κάτι το συγκεκριμένο από μέρους του Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία. Ευχαριστούμε κυρία Τρανταφυλλίδη. Και τώρα από τις κάτω χώρες, από την κάτω βουλή της χώρας, ο κύριος Βίμερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω τις ε, ερωτήσεις μου, οι οποίες νομίζω θα ήθελα απάντηση από την ε, εκπρόσωπο της Επιτροπής. Γιατί αντί να ορίζουμε το όριο στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις υπό τους 250 ε, εργαζομένους, γιατί να μην ορίσουμε τα όρια ως προς τον όγκο των ε, δεδομένων που την χάνουν επεξεργασίες. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι όλοι θέλουν να προστατεύσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ανεξαρτήτως του μεγέθους της, μία επιχείρηση, εφόσον είναι στην, ε, στο χώρο της ε, κατεργασίας δεδομένων, μπορεί να αναλάβανε την επεξεργασία δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών. Γιατί λοιπόν να μην επιλέξουμε μια διαφορετική γραμμή εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, εμείς σας ευχαριστούμε και πάλι από την Πολωνική Βουλή ο κύριος Αντρέ Γκαλατσεύσκη για δύο λεπτά. E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά την παρέμβαση της συναδέλφου από την Επιτροπή Δικαιοσύνης, πρέπει να πω ότι εξετάζουμε τις δύο νομοθετικές προτάσεις και έχουμε συνομιλίες ε, με εμπειρογνώμονες για το θέμα αυτό. Ήθελα και εγώ λοιπόν μετά την παρέμβαση της αδέλφου μου να προσθέσω δύο σχόλια. Ήταν εύστοχε οι παρατηρήσει τη Ιταλίδα συναδέλφου, τη κυρία Αλεγκρίνη, για την μονοπεθυντική θηρίδα, το one-stop shop. Εδώ το τι εκδοχή θα προβλεφθεί είναι πολύ σημαντικό και θεωρούμε ότι δύσκολο θα είναι να εφαρμοστεί το δικαίωμα στη λύθη. Στην σημερινή πραγματικότητα οι πληροφορίες ε, μεταδίδονται και αποστέλλονται με τρόπο που ελέγχεται ελάχιστα. Θα είναι λοιπόν λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη πιστεύω. Τέλος, να πω ότι οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό πολλές φορές δεν έχουν ειδική μεταχείριση για τα ευαίσθητα δεδομένα που έχουν σχέση με την υγεία. Αυτά πολλές φορές μεταφέρονται διακρίτως και δεν προβλέπεται ειδική προστασία για τα θέματα αυτά. Θα πρότεινα λοιπόν στη Γενική Διευθύντρια και για τι δύο νομοθετικέ προτάσεις να φροντίσει να λάβει αυτά τα στοιχεία υπόψη και να γίνουν οι απαραίτητε τροποποιήσεις στα κείμενα. Ή έστω να προβλεφθεί η διευκρίνησή του με κατεξουσιοδότηση πράξη. Πρόεδρος. Ακούσαμε μια σειρά ερωτήσεων. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να τηρήσει κανείς το χρόνο του αυστηρά. Έχουμε όμως μερικά λεπτά στη διάθεσή μας ακόμη για να ακούσουμε τις απαντήσεις από την έδρα. Θα πρότεινα να ακούσουμε με την ίδια σειρά τις παρεμβάσεις και έτσι τρία-τέσσερα λεπτά μόνο παρακαλώ για να απαντήσει ο καθένας ε, εκ των ομιλητών εκ μέρους της έδρας. Ο κύριος Νικολάου παρακαλώ. Πάρα Θα αρχίσω από το, την πρώτη ερώτηση που έχει τεθεί από τη ΣΕΑΡΦ από την Ισπανία για το ζήτημα της εμπιστοσύνης των πολιτών. Σίγουρα μια αποτελεσματική, σαφής θα έλεγα νομοθεσία η οποία θα μπορεί να εμπνεύσει ασφάλεια στους πολίτες μέσα από τις διατάξεις της και τις ρυθμίσεις ειδικότερα πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κατοχυρώνονται μια σειρά από δικαιώματα μέσα στον κανονισμό όπως είναι η πρόσβαση, όπως είναι η διόρθωση, όπως είναι η διαγραφή λήθης παρά το γεγονός ότι πράγματι υπάρχουν δυσκολίες και προβληματισμός στο κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η δυνατότητα αλλά η τεχνολογία είναι τέτοια που νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει και λύση σε αυτό το ζήτημα να αναγνωριστεί το δικαίωμα διαγραφής είναι ένα σημαντικό ζήτημα όπως επίσης και το δικαίωμα της μεταφοράς είναι το δικαίωμα της προσφυγής κατά της αρχής ελέγχου ή ακόμα και το δικαίωμα της προσφυγής κατά του υπευθύνου επεξεργασίας Αυτά είναι δικαιώματα τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν στον πολίτη και ο πολίτη μέσα από αυτέ τι διαδικασίε να μπορεί να δώσει εμπιστοσύνη στην εφαρμογή αυτού του κανονισμού που όταν μιλούμε για έναν κανονισμό ο οποίο θα εφαρμοστεί ε, ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη-μέλη και στα 27. Ε, τώρα, για το ζήτημα που έχει θέσει ο κύριος Τριανταφυλλίδης, γιατί η αναθεώρηση καθυστερεί ε, και ότι είναι αναγκαία, θα έλεγα το εξή. Όταν μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα και όταν επιχειρείται η προστασία μέσω νομοθεσίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ίσως από την πιο δύσκολη νομοθετική εργασία που μπορεί να, να επιτελέσει έναν, ε, μια, έναν κατεξουσιοδοτημένο όργανο. Γι' αυτό τον λόγο και όταν ειδικότερα αυτά τα δικαιώματα επιχειρείς την ίδια ώρα που τα κατοχυρώνεις επιχειρείς και να τα περιορίσεις για σκοπούς ισορροπίας η αναζήτηση αυτής της ισορροπίας επιβάλλει να υπάρξει αυτός ο διάλογος που γίνεται σήμερα, επιβάλλει να υπάρξει μια επαρκής, θα έλεγα, συζήτηση για να φτάσουμε στο σημείο το οποίο χρειάζεται για να δώσουμε μια αποτελεσματική λύση ε, νομοθετική στου ε, πολίτες μας. Δεν νομίζω να υπάρχει ουσιαστική καθυστέρηση. Είναι, επηρεάζονται ξεκάθαρα σημαντικά συμφέροντα από αυτή τη ρύθμιση, από αυτή την νομοθεσία είναι αυτά που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση που χρειαζόμαστε. Τώρα για την κατεξουσιώδη συμπράξη, σίγουρα είναι υπερβολικό ο αριθμό των κατεξουσιώδη συμπράξεων και εμεί ω Εθνικό Κοινοβούλιο ε, Κυπριακή Βουλή έχουμε εντοποθετηθεί ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ένας προβληματισμός εκ νέου, μια αναθεώρηση ε, της ε, ρύθμισης αυτής, αλλά και την ίδια ώρα πιστεύω ότι εκεί που θα δοθεί κατεξουσιώδηση ε, πράξη ε, το δικαίωμα αυτό πρέπει να περιορίζεται εντός των ρυθμίσεων του κανονισμού. Δεν μπορούμε με κατεξουδότηση πράξης να υπερβαίνουμε τον κανονισμό. Κατά τη δική, ε, κάτι για μας τους νομικούς αυτό θα ήταν ultravirus του κανονισμού και οι πράξεις θα ήταν χωρίς εξουσιοδότηση ουσιαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. ευχαριστώ κύριε Νικολάου. Ο κύριος Υπουργός, παρακαλώ. Εκεί που έμεινε ο κύριος Νικολάου όσον αφορά τις κατεξουσιοδότης πράξη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και προβληματίζει, μπορώ να πω, όλα τα κράτη-μέλη. Και λαμβάνοντας, αφουγκράζοντας αυτές τις ανησυχίες των κρατών μελών, το είχαμε θέσει σαν θέμα συζήτηση στο άτυπο συμβούλιο των Ιούλιο, το 23-24 Ιουλίου που έγινε στην Λευκοσία. Η καθοδήγηση που είχε δοθεί από το Συμβούλιο είναι ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι να μειωθούν αυτές οι κατεξουσιοδότη πράξεις. Ήταν η γενική τοποθέτηση των κρατών μελών ότι είναι υπερβολικός ο αριθμός. Θα κάνω μια γενική τοποθέτηση. Όσον αφορά το δικαίωμα λήθης, ε, το άρθρο 17, υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες αποτελεί όμως ένα πρώτο βήμα για τον έλεγχο από το ίδιο το υποκείμενο. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε χρόνο να τελειώσουμε με καλή θέληση όλοι οι εμπλεκόμενοι. Νομίζω ότι δεν είναι σοβαρό θέμα και πρέπει να επιληθεί αυτό και θα επιληθεί. Ε, όσον αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Τριανταφυλλίδη γιατί κανονισμό και γιατί ε, οδηγία, γιατί να το διαχωρίσουμε. Όπως έχω αναφέρει και στην ομιλία μου, αυτά τα δύο ε, μέτρα προχωρούν μαζί. Και έχει εξεταστεί ένας αρκετά μεγάλος, μπορώ να πω, άρθρων, αριθμός άρθρων ε, το, τους τελευταίους δύο, μισή μήνες. Όπως και αρχίσαν και εξετάζονται και έχουν εξεταστεί τα πρώτα άρθρα της οδηγίας. Όπως ήταν γενική διαπίστωση ότι η υπάρχουσα νομοθεσία ε, βασικά είχε δημιουργήσει 27 εθνικές νομοθεσίες και είδαμε ότι δεν ήταν αποτελεσματική. Γι' αυτό η αντικατάσταση της οδηγίας με έναν κανονισμό που εκ της του αποτελεί ένα λιγότερο νομοθετικό, ελαστικό νομοθετικών εργαλείο και δεν επιτρέπει στα κράτη-μέλη τη θέσπιση ουσιαστικών παρεκκλήσεων σε εθνικό επίπεδο. Ε, σίγουρα προβλήματα υπάρχουν, αλλά είμαστε εδώ που με συνεργασία όλων, όλων των εμπλεκομένων, δεν είναι εκτός από το Ευρωκοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο, έχουμε να συζητήσουμε και με τις επιχειρήσεις. Αυτόν κάνει η Προεδρία, γιατί πρέπει να, πάρουμε, να ενημερώσουμε και να πάρουμε απόψεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καθυστέρηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό νομοθέτημα για να το διαβούμε γρήγορα γρήγορα. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να παραδώσουμε έναν ποιοτικό έργο στην επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία, ούτως ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Όσον αφορά τον την οδηγία, ναι, επειδή αυτό θα αφορά θέσπιση κανόνων προστασία των προσωπικών σε εθνικό επίπεδο στον τομέα τη αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει, πρέπει να υπάρχει κάποια ελαστικότητα εδώ, πιστεύω, όσον αφορά τι αρχέ επιβολή του νόμου, τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσουμε να, επιτεχ... να, να, να εύρουμε το ισοζύγιο μεταξύ των ατομικών δικαιωμάτων, των ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την, αποτελεσματική, την αποτελεσματικότητα της αρχής των αρχών επιβολής του νόμου. Ε, νομίζω κύριε Πρόεδρε, ε, νομίζω, κύριε Πρόεδρε έχω κάνει μια γενική τοποθέτηση. Δεν ξέρω αν έχει διαφύγει οτιδήποτε. Εκείνο που θέλω να, σαν, σαν τελευταία τοποθέτηση είναι η αυτόν το θέμα είναι η απαραίτητη συνεργασία όλων. Στενή συνεργασία Ευρωκοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου. Μόνο έτσι θα πετύχουμε. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Και παρακαλώ τώρα την κυρία Λεμπάιλ, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να λάβει τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις ε, ερωτήσεις που δεν ε, απάντησαν, δεν έθιξαν οι προηγούμενοι ομιλητέ. Αναφερθήκατε στην επικουρικότητα καταρχάς. Για την επικουρικότητα, εν συντομία θα ήθελα να πω ότι το άρθρο 6 του χάρτη καθιστά υποχρεωτική την εξασφάλιση εφάμιλου επίπεδου προστασία των δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ είναι η αναφορά στο άρθρο 16, νομική βάση δηλαδή, από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αρχή της επικουρικότητας της προτάσεις μας. Και πάλι για την κυρία Αγγελίνη, είπατε ότι λυπάστε που ο πολίτης δεν μπορεί πλέον να στραφεί στις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της πατρίδας του. Θα ήθελα να επισημάνω όμως ότι αυτό δεν αληθεύει. Πάντοτε ο πολίτης θα μπορεί να προσφύγει στην αρχή προσωπικών δεδομένων της πατρίδας του. Οι εθνικές αυτές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα έχουν επικοινωνία, επαφή με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έχει επιληφθεί της ε, υπόθεσης ενδεχομένως αλλά εμείς μεριμνούμε με ιδιαίτερη προσοχή να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα, γιατί ήταν πολύ σημαντικό για μα το να μπορεί ο πολίτης ή αντίστροφα η εθνική αρχή προσωπικών δεδομένων να παραμένει κοντά στον πολίτη τη. Η άλλη ερώτηση που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιλογή των 250 εργαζομένων για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτή η επιλογή οφείλεται στο, βασική, στο βασικό ορισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση του τι συνιστά μικρομεσαία επιχείρηση. Ένας απλός ορισμός, αποδεκτός από τους πάντες και ο οποίος ορισμός αποτελεί την βάση μια σειρά μέτρων και ε, νομοθετημάτων. Ως εκ τούτου λοιπόν και επί της αρχής παλάσσονται από τις προϋποθέσεις ως προς την τεκμηρίωση και λοιπές προϋποθέσεις στις οποίες υπάγονται άλλες επιχειρήσεις και τι πάλι υποχρεούνται να τηρούν την ίδια νομοθεσία. Ωστόσο, έχουμε, έχουμε εκτιμήσει μάλλον ένα παράγοντα κινδύνου στην υπόθεση αυτή και όπως πολύ σωστά επισημάνατε και εσείς, μπορεί μια πολύ μικρή μικρομεσαία επιχείρηση να διαχειρίζεται γιατί αυτή θα είναι η εξειδικευσή της, ο τομέας της, να διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα και μάλιστα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ε, σε τεράστιους όγκους. Γι' αυτό λοιπόν στην νομοθεσία εισάγουμε μια θα έλεγα εξαίρεση, η οποία λέει ότι αυτές οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ε, χειρίζονται, επεξεργάζονται δεδομένα, προσωπικά δεδομένα, παραμένουν υπάγονται δηλαδή πάντα στις προϋποθέσεις προστασίας, στις ασφαλιστικές δικλίδες που έχουμε όπως αξιολόγηση συνέπειών, στέλεχος προστασίας προσωπικών δεδομένων, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί η βασική δουλειά τους είναι η προστασία των δεδομένων. Για τον κύριο Κάλιτς, αναφερθήκατε στην ασαφή διατύπωση ε, κακή διατύπωση άκουσα εγώ από τη διερμηνία, σαφή διατύπωση εν πάση περιπτώσει ε, για το κείμενο των άρθρων. Προφανώς πρέπει να αναθεωρήσουμε και να καταστήσουμε πιο σαφή τη διατύπωση των άρθρων αυτών. Αυτή είναι και η προσπάθεια με το συνομοθέτη μας στην οποία αποδιόμαστε, να καθιστούμε δηλαδή δυνατόν για οποιονδήποτε θέλει να διαβάσει την νομοθεσία αυτή, για όποιον θέλει να διαγνώσει τη σκοτεινή πλευρά των όσων προτείνουμε, να είναι πιο ευχερής, πιο ευανάγνωστο ουσιαστικά το κείμενο, πιο ευχερής η ανάγνωση. Να είναι προσβάσιμο σε περισσότερους ανθρώπους. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη για διευκρίνηση της ε, διατύπωσης και βεβαίως δεχόμαστε τις υποδείξεις που έχετε ενδεχομένως να κάνετε. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα που έθιξε επίσης η κυρία Αλεγκρίνη. Έχουμε όντως προσπαθήσει να καταστήσουμε πιο απλή την ε, προστασία, διατηρώντας όμως την επίπεδό της. Άρα, όταν μπορεί κανείς να μεταφέρει δεδομένα, προσωπικά δεδομένα σε, τρίτα, σε τρίτη χώρα. Καταρχάς θα έχουμε τη διαδικασία της προσαρμογής που έχει ήδη ξεκινήσει. Θα έχουμε μια απλουστευμένη μορφή για επιχειρήσεις και κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν τους ειδικού κανόνες που για, αυτούς, για αυτές και βεβαίως θα έχουμε και τις εγγυήσεις, που τις συμβατικές εγγυήσεις Άρα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα, θα έλεγα, δυνατοτήτων για μεταφορά δεδομένων, ταυτόχρονα όμως διατηρώντας, και αυτό είναι το ουσιαστικό, ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λεμπάια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νικολάου, κύριε Λουκά. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο Σούλτς, ο οποίος ε, ήρθε στο πρώτο τμήμα της ε, συνεδρίας. Ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν το λόγο. Μερικές φορές δυσκολευόμεθα να, να τηρούμε το χρόνο μας, τα χρονικά μας όρια, αλλά τα καταφέραμε αυτή τη φορά. Καταφέραμε εγκαίρως να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε το δεύτερο κομμάτι της σημερινής μας συνεδρίασης, του οποίου θα ηγηθεί ο κύριος Γιάνν Φιλιπ Άλμπρεχτ, αρμόδιος ε, για την έκθεση σχετική με τις ρυθμίσεις ε, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων από την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και ε, Εσωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα γίνει αλλαγή προσώπων εδώ στην έδρα του Προέδρου και το δεύτερο τμήμα της συνεδριάσεως θα ε, πάει μέχρι τις 12.30. Θα διακόψουμε μετά για το μεσημεριανό μας. Εγώ σας υπενθυμίζω ότι η Αντιπρόεδρος κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ, η οποία είναι και αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης και πολιτικών ελευθεριών επίτροπος, θα ε, κηρύξει την έναρξη του απογευματινού τμήματος της ε, συνεδριάσεως στις 3 ακριβώς το απόγευμα. Σας ευχαριστώ και πάλι και αφήνω τη θέση μου για τον επόμενο πρόεδρο στην έδρα. Dear ladies and gentlemen, I would like. Κυρίες και κύριοι. Come everybody. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης αυτής της μικτής διάκοινοβουλευτική καλύτερα συνεδρίασης. Ο χρόνο βέβαια προχωράει γοργά και πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να σταματήσουμε στις 12.30. Ο, ο μιλητής λέει 2.30. Εν πάση περιπτώσει, στις 12.30 θα πρέπει να σταματήσουμε. Είπε ο πρόεδρος μας ότι έχουμε διερμηνία. Καλείστε οι πάντες να μιλάτε τη γλώσσα σας, λέει ο, ομιλητής. Έχουμε εδώ διακεκριμένους ομιλητές στο δεύτερο αυτό τμήμα που αφορά την ε, εναρμονισμένη και ενισχυμένη προστασία προσωπικών δεδομένων, δικαιώματα και αρχές για έναν αλληλοσυνδεόμενο κόσμο. Ας περιορίσουμε λοιπόν τις ομιλίες μας Έχουμε αρκετούς ομιλητές, όπως είπα, και σημαντικές παρεμβάσεις. Αυτό δεν θέλω να μακρηγορήσω εγώ ως εισηγητής. Έχω αρκετές φορές την ευκαιρία να μιλάω. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους προσκεκλημένους στα δεξιά μου, στα δικά σας αριστερά. Είναι η κυρία Μαριέτα Καραμαντλή, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ε, Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Την καλωσορίζω. Ο Γκέριτ Χόρνουγκ από το Πανεπιστήμιο του ΠΑΣΑΟ. Στα αριστερά μου ο Ζων Γκονί, ε, διευθυντής θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων ιδιωτικού βίου της ε, Microsoft Europe. δίπλα του η κυρία Νούρια Ροδρίγκες από την Ευρωπαϊκή από την οργάνωση, Ευρωπαϊκή Καταναλωτών ε, στο, από την νομική υπηρεσία τους και ο κύριος Σάιμον Ντέιβις ε, στην άκρη από το London School of Economics. Ξεκινούμε λοιπόν ε, με ένα δεκάλεπτο για τον καθένα και την κυρία Μαριέτα Καραμανλή πρώτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τις κυρίες και κύριοι η μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων ε, και η πρόταση οδηγίες τον περασμένο Γενάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν μεγάλη σημασία. Έχει μια ιδιαιτερότητα το θέμα αυτό, διότι από τη μια αγγίζουμε τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, απ' την άλλη έχουμε και τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις. Το δικαίωμα δηλαδή της προστασίας των δεδομένων, σας υπενθυμίζω, εντάσσεται στο άρθρο 8 της Χάρτας των Ευρωπαϊκών Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στη η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε σε αυτό το θέμα. Και, λοιπόν, το ψηφιακό θέμα, όπως αναφέρθηκε, έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και δουλεύουμε και το ρυθμιστικό πλαίσιο των χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσαρμοστούν Έχουμε μια έκρηξη των κοινωνικών δικτύων, των οργανισμών, υπάρχει μια γενικοποίηση. Έχουμε να κάνουμε με την, το χειρισμό όλων αυτών των δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει καταθέσει μια πρόταση κανονισμού. Ε, δεν είναι κάτι το καινούριο. Έχει όμως μεγάλες συνέπειες όσον αφορά την αρμόνιση των δικαιωμάτων. Ο κανονισμός, υπενθυμίζω, θα εφαρμοστεί άμεσα και δεν θα, έχει, δεν θα ισχύει αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να περάσουμε σε αποτελεσματικότητα, μια εναρμόνιση και θα έλεγα ότι αυτή η εξέλιξη ε, δεν, σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν ρίσκους όσον αφορά να υπάρχουν ε, ανισότητες όσον αφορά τις ε, νομοθεσίες των χωρών μελών. Θα πρέπει κατά με λοιπόν καταρχήν να υπογραμμίσουμε ότι η πρόταση κανονισμού σημαίνει μια πρόοδο, θετικά αυτά, μπορούμε να μιλούμε για μια πρόθεση δικαιωμα... της προστασίας των δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Αυτά είναι πολύ θετικά και τα περιμέναμε. Έχουμε την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου, έχουμε αναφορές όπως τα δικαιώματα στη Υπάρχουν παρόλα αυτά πολλά ερωτήματα όσον αφορά την ε, δυνατότητα να εφαρμόσει κανείς ένα κάτι τέτοιο. Αυτό το δικαίωμα στη ε, προβλέπεται στο άρθρο 17, στην πρόταση κανονισμού. Είναι λοιπόν το άτομο το οποίο θα μπορέσει να ζητήσει την ε, διαγραφή δεδομένων. Υπάρχει αυτή η πρόθεση. Επίσης υπάρχει το θέμα της προστασίας των δικαιωμένων για ένα άτομο τα οποία έχουν ε, δοθεί όταν ένα άτομο ήταν παιδί, ανήλικος. Και αν θελήσει λοιπόν ένα άτομο αργότερα μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή του δικαιώματος τη λύθη. Αυτές οι, προ... οι προτάσεις λοιπόν δημιουργούν προσδοκίες και ο νομοθέτης ο Ευρωπαίος θα πρέπει να απαντήσει. Εδώ έχουμε να κάνουμε και την ικανότητα του να δημιουργήσει ένα δικαίωμα λύθης το οποίο είναι εφαρμόσιμο κάτι το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί, δεν είναι ξεκάθαρο σήμερα. είχαμε την γνωμοδότηση 7 Μαρτίου του 2012 για όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας σαφής ε, ορισμός όσον αφορά το άρθρο 17. Τώρα για την ε, μεταφορά δεδομένων. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να δίνεται μια κόπια στον ε, υπεύθυνο και μετά να γίνεται χρήση. Αυτό το δικαίωμα είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να διευκρινιστεί. Το κείμενο θα πρέπει να αφορά μόνο ε, τη χρήση δεδομένων, να διασαφηνίζει ακριβώς πώς θα γίνει η χρήση στα πλαίσια των δικαιωμάτων όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία κλπ. Είναι πάρα πολλά αυτά τα ερωτήματα και όλα αυτά θα πρέπει να, τα, να μας προβληματίσουν. Τώρα, για την ενίσχυση τη, πολύ ουσιαστική των υπαρχόντων δικαιωμάτων και αυτό σημαίνει μια μεγάλη πρόοδο, μίζωνα. Ε, έχουμε να κάνουμε τη συνένεση, το δικαίωμα ενημέρωση του, ε, του πρόσωπου το οποίο αφορά τη δυνατότητα του ατόμου να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και επίση το δικαίωμα να αρνείται να γίνεται χρήση δεδομένων. Όλα αυτά μα δίνουν τη δυνατότητα να πετύχουμε μια ισορροπία στον κανονισμό υπέρ του Ευρωπαίου πολίτη για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων. Ο αρμόδιο των δεδομένων θα πρέπει να έχει μια, μια επαφή άμεση και απλή με το πρόσωπο το οποίο αφορά θα πρέπει να ενισχυθεί η προστασία του και όταν θα πρέπει να περάσουν σε κάποιον άλλο άτομο θα πρέπει να να απαγορεύεται να γίνει χρήση των δομέτων αν δεν υπάρχει συνένεση του προσώπου των οποίων αφορούν. Υπάρχει το θέμα φυσικά της παθητικής συνένεσης ή σιωπήλας. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη συνένεση του προσώπου. Έχουμε τώρα την περίπτωση των δυνατότητας δεδομένων τα οποία μπορεί να δίδονται από ένα γονέα το, θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα είναι πιο αυστηρά όσο αφορά τη διάδοση των δεδομένων και στη συνέχεια θα υπάρχει το θέμα της εγγύησης των δικαιωμάτων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την ευθύνη αυτού που είναι υπεύθυνο για τα δεδομένα. Θα πρέπει ε, να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί να γίνει κατάχρηση όσον αφορά την προστασία αυτών των δεδομένων. Υπάρχει επίσης ε, μια, ένα συγκεντρωτισμό όσον αφορά τον έλεγχο. Το, η πρόταση κανονισμού ε, δημιουργεί σημαντικές αλλαγές όσον αφορά το άρθρο 12. Έχουμε το δικαίωμα ενημέρωσης των ατόμων σε σχέση με τη χρήση των δεδομένων από τον υπεύθυνο. Υπάρχουν οι γενικές συνθήκες όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων. Η τώρα το θέμα της διάρκειας όσον αφορά τις ε, ε, αποθήκευση των δεδομένων, ε, το θέμα που έχει να κάνει από πού έρχονται τα δεδομένα, αν έχουν γίνει άμεσα ή όχι σε σχέση με το πρόσωπο το οποίο αναφορούν. Επίσης το σχέδιο κανονισμού ζητά από τον υπεύθυνο να προστατεύσει αυτά τα δεδομένα, να υπάρχει διαφάνεια και να είναι εύκολα προσβάσιμα. Επίσης θα πρέπει να γίνει σωστή κατάρτιση των πολιτών, εφαρμοστούν οι βέλτιστε πρακτικέ στα πλαίσια των δικήσεων. Χρειάζεται να γίνεται έλεγχο από τι εθνικέ αρχέ και έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι απαραίτητο όταν μιλάμε για αυτό το νέο δικαίωμα. Και φυσικά θα πρέπει να προγραμμιστούν ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω πρόοδοι. Έλεγχο σε εθνικό επίπεδο. Απ' την άλλη έχουμε το θέμα τη ενίσχυση και εναρμόνιση, ούτω ώστε να υπάρχει ε, και η εγγύηση και η ανεξαρτησία στη χρήση των δεδομένων. Επίσης, οι αρμοδιότητες τώρα των εθνικών αρχών, όπου θα πρέπει έχουμε να κάνουμε με την, το χώρο της κύριας εγκατάστασης, θα πρέπει να ξέρουμε να γίνεται κατανοητό ότι μπορεί κανείς να αναλάβει και να βοηθηθούν οι όποιες ε, ε, επιφυλάξεις. Έχουμε να κάνουμε τις ε, αρχές οι οποίες είναι πιλωτικές, οι εθνικές, θα πρέπει να έχουν τις αρμοδιότητες για να μπορέσουν φέρει πει να δεχθούν μια, ένα παράπονο και να μπορέσουν να το εκπαιρεώσουν. Θα υπάρξει μια αρχή σε εθνικό επίπεδο που θα κινηθεί πολιτικά και να περάσει πέσει και σε κυρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει αξιολόγηση, να αξιολογήσει όλες τις εναλλακτικέ προτάσεις για να προστατεύσει τον πολίτη. Η πρόταση λοιπόν, ε, η αρχική ίσως να μην είναι πολύ ικανοποιητική. Και πριν να κλείσω κύριε συνάδελφοι, δύο σημεία τα οποία θα πρέπει να υπογραμμίσουμε σε σχέση με την εμφάνιση των δικαιωμάτων σε αναρμονισμένο επίπεδο. Το κείμενο δίνει τη δυνατότητα ε, ε, σφυγή όσον αφορά στις ε, ε, ή τις εκτελεστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν πολλές ασάφειες, θα πρέπει να τις ξαναδούμε στα πλαίσια του κανονισμού. Επίσης να πω ότι λυπάμαι που ότι το νομοθετικό πακέτο είναι κατακαιρματισμένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατέθεσε δύο κείμενα σε σχέση με την οδηγία του 92 και σε σχέση με την νομοθεσία ε, πλαίσιο του 98. Όλα αυτά έχουν δεχθεί κριτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα δεδομένα, η μεταμόρφωση θα μας δώσει δυνατότητα να προχωρήσουμε στα δύο κείμενα. Τα πράγματα όμως έχουν υποκαριστεί. Είναι λοιπόν επίγον να δούμε αυτά τα δύο θέματα. Και το τελευταίο σε οποίο φυσώ την προσοχή. Αν αυτά τα, αυτά τα μέσα που έχουμε θα πρέπει θα πρέπει να τα δούμε και θα μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να τα αναθεωρήσουμε. Θα υπάρχει μια συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ξαναδουλέψει κανείς πάνω σε αυτά τα θέματα. Υπάρχουν σίγουρα και άλλα ουσιάδη θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δουλέψει κανείς στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Uh, Οι διερμηνείς πρέπει να αναπτύξουν ταχύτητα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να παίρνει κανείς το λόγο πρώτη φορά, αλλά καλό θα ήταν να μιλάμε με κάπως ε, αργότερο ρυθμό για να προλαβαίνουμε να τα μεταφράζουμε κιόλας. Ο κύριος Χόνουγκ τώρα υπεύθυνο για την νομική διάσταση της πληροφορικής, ερευνητή που σχολίασε από τους πρώτους της προτάσει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Πανεπιστήμιο του Πάσαου. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ και εγώ έχω δυστυχώ την κακή θύμη ότι είμαι πολύ γρήγορος ομιλητή. Ευχαριστώ λοιπόν όλου του παρεμβαίνοντε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι προτάσει τη. Νομίζω ότι τι οφείλουμε ευχαριστίε ακριβώ γιατί είναι αξιόλογε οι ιδέε ε, στα κείμενα. Αλλά στο επόμενο δεκάλεπτο θα ήθελα να επικεντρωθώ στα σημεία όπου θα μπορούσαν να επιφερθούν βελτιώσει στα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων. Πρώτα απ' όλα για τα δικαιώματα δεν θα επικεντρωθώ στα ισχύοντα. Νομίζω ότι ήδη προστατεύονται επαρκώ. Ήθελα να σταθώ στα νέα σημεία. Η κατάρτιση προφίλ, ένα νέο στοιχείο που νομίζω ότι είναι βήμα πρόοδου, δηλαδή η συλλογή ενό μεγάλου έγκου, όγκου δεδομένων για ένα συγκεκριμένο άτομο, ένα συγκεκριμένο πολίτη. Αυτό το νέο στοιχείο δεν είναι τελικά και τόσο καινούργιο, γιατί το άρθρο 20 περιορίζει τα μέτρα αυτά κατάρτιση προφίλ μόνο στα εκτονιστέρων ε, μέτρα που μπορεί να ε, λυθούν, όχι στην ίδια την κατάρτιση του προφίλ. Η κατάρτιση προφίλ αυτή αυτή θεωρώ ότι είναι κάπως προβληματική έννοια. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι οι αμφιλεγόμενοι περιορισμοί για τις περιπτώσεις ανισορροπίας μεταξύ του ατόμου για το οποίο σου λέγονται τα δεδομένα και του ελεγχτή από την άλλη. Η τη ισορροπία νομίζω ότι είναι ένα βήμα προόδου και θα πρέπει να διευκρινιστεί στην πρόταση ποιε περιπτώσει ανισορροπία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Ποιε θεωρείται ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν η αιτιολογική σκέψη 34 αναφέρεται στο χώρο εργασία, αλλά νομίζω και σε άλλε περιπτώσει μονοπωλίου θα πρέπει να τα σκεφτούμε ω περιπτώσει. Επίσης, οι χρήστε θα μπορούσαν να υποφεληθούν από τα λεγόμενα patch της εξελιγμένες μορφές τεχνολογίας. Εδώ δεν υπάρχει όμω κάποια δεσμευτική δήλωση ω προ το σχεδιασμό των τεχνολογιών και δεν υπάρχουν και γενικέ αρχέ για την επεξεργασία των δεδομένων μέσα από τα τεχνολογικά μέσα. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν κάποια ευθυγράμμιση, κάποιο συντονισμό. Ε, επίσης, οι σφραγίδες και τα σήματα της ε, συλλογή δεδομένων είναι και αυτό σημαντικό. Ο κανονισμό όμω δεν θα πρέπει απλώ τα ασαφή καθήκοντα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των Κατώμελών μελών να τα διευκρινίζει, να τα ενθαρρύνει μάλλον απλώ, θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένε διατάξει για το ποιο θα μπορεί να ε, επιφέρει, να επιβάλλει, να επισυνάπτει μάλλον αυτές τις σφραγίδες, ποια θα είναι τα ισχύοντα κριτήρια και ποιες οι νομικές συνέπειες αυτών των σημάτων και σφραγίδων που θα επιφέρονται στα, στην περίπτωση της προστασίας δεδομένων. Όλα αυτά συζητώνται εντατικώς προκειμένου να υπάρξει εθνική νομοθεσία τη Γερμανία τουλάχιστον και η αρμόδια Γερμανική Επιτροπή δεν πέτυχε να καταλήξει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν συμφώνησαν τα μέλη του Κοινοβουλίου στη Γερμανία μεταξύ του. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσω με πολύ δυσκολία βέβαια να βρει κάποια λύση εδώ, αλλά είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί αυτό στην πρόταση. Επίση για τα προτινόμενα και τα ισχύοντα δικαιώματα, ένα θέμα είναι αυτό τη επιβολή του νόμου, το ρόλο των διοκτικών αρχών. Το να υπάρξουν μηχανισμοί πραγματική επιβολή είναι πολύ σημαντικό γιατί μόνο έτσι τα μέτρα θα γίνουν πραγματικά ε, πράξη. Είναι λοιπόν σημαντικοί οι μηχανισμοί. Ε, εδώ η πρόταση για το μηχανισμό συνεκτικότητας είναι ήδη προβληματική, διότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη βεβαίω να παρέχουν πλήρη ανεξαρτησία στι ελεγκτικέ αρχέ σε εθνικό επίπεδο, αλλά ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα οργανισμό, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να έχει τον τελικό λόγο ώστε να διασφαλίζεται η πλήρη ανεξαρτησία τη επεξεργασία των δεδομένων. Αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί μέσα στη διαδικασία μεταρρύθμιση. Τώρα, για τα νέα δικαιώματα, δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα για τη φορητότητα, δηλαδή τη δυνατότητα μεταφορά των δεδομένων. Είναι σημαντικό αυτό, να μπορεί να μεταφέρονται τα δεδομένα από τον ένα ελεγκτή στον άλλο. Αυτό είναι ένα βήμα πρόοδου, διότι έτσι θα μπορούν να προβλεφθούν και να προληφθούν οι δυσμενείς ε, για τους πολίτε τα άτομα για τα οποία συλλέγονται δεδομένα. Αλλά ας πούμε ότι κάποιος ε, μπορεί να πάρει τα δεδομένα του και να τα πάρει από ένα κοινωνικό δίκτυο, να τα πάει σε ένα άλλο, αλλά μετά να μην τα ξαναπάει πίσω. Αυτό σημαίνει ότι τελικά το δικαίωμα θα πέσει σε αχρηστία. Εδώ δεν έχουμε απλώ ζητήματα προστασία δεδομένων σε κάθε περίπτωση. Τώρα για το διαβόητο δικαίωμα στη λύθη, δικαίωμα δηλαδή διαγραφή. Εδώ Νομίζω ε, χρειάζονται περισσότερε λεπτομέρειε από όσα ήδη προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα είναι αν θα δημοσιεύονται τα δεδομένα ή αν θα μπορούν να μεταδοθούν ή αν θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενο εκ των υστέρων. Ο ελεγκτή θα πρέπει να ενημερώνει όλου του ελεγκτέ όταν γίνεται η διαγραφή. Δηλαδή, εάν και άλλοι έχουν ε, ασκήσει επεξεργασία στα ίδια δεδομένα, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Πώ θα γίνεται όμω αυτό. Ο ελεγκτή έχει δημοσιοποιήσει, α πούμε, τα δεδομένα. Αυτό δεν το γνωρίζουν αναγκαστικά τα υπόλοιπα μέρη. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει και αυτή η έννοια της δημοσίευσης των δεδομένων. Έπειτα η υποχρέωση ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, αυτούς δηλαδή από τους οποίους προέρχονται τα δικαιώματα. Εδώ θα πρέπει να εξευρεθεί η ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και των αναγκών δημοσίευσης χωρί να τίθεται να αμφιβόλω η προστασία των δεδομένων. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να προσπαθεί να επιλύσει το ουσιώδε πρόβλημα των διαδικαστικών καθηκόντων. Νομίζω το πραγματικό πρόβλημα εντοπίζεται στο άρθρο 80, διότι εκεί προβλέπονται εξαιρέσει και παρεκκλήσει για τα κράτη-μέλη ω προ την ελευθερία του λόγου και την ελευθεροτυπία. Όμω, δεν μπορεί κανεί να έχει και τα δύο. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ευρωπαϊκό δικαίωμα διαγραφή ή δικαίωμα στη λύθη και από την άλλη εθνικέ ρυθμίσει για την ελευθεροτυπία και την ε, ελευθερία του λόγου. Διότι ακριβώς εκεί ε, δίνεται στους ελεγκτές το δικαίωμα να άρουν το δικαίωμα λήθη, το δικαίωμα διαγραφής. Είναι αντιφατικά αυτά μεταξύ τους. Έπειτα για τις αρχές ε, που υπόκεινται στην κατάρτιση των δικαιωμάτων. Υπάρχει εδώ μια οδηγία που ήδη ισχύει και θα πρέπει να εξεύγουν μια κατάλληλη νομική βάση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο το, η δυνατότητα της ε, εφαρμοσιμότητας των μέτρων. Κάποια στιγμή τα δεδομένα μπορεί να είναι παροχημένα, να μην είναι πλέον σημαντικά. Θα πρέπει οι ελεγκτές να μπορούν να τα επεξεργαστούν όπως δει. Θα πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν για το πλαίσιο χρήση των δεδομένων, όχι για τη δυνατότητα ε, υλοποιησιμότητας. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε εάν για το δημόσιο συμφέρον βάσει του άρθρου 6 είναι χρήσιμη η επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ιδιαίτερα η έννοια του δημόσιου συμφέροντος. Στο άρθρο 6.3 αναφέρονται και ε, περαιτέρω προϋποθέσεις για τις επιμέρους ανάγκες των κρατών που μπορεί να προκύψουν. Τι εννοούμε όμω ακριβώ με το δημόσιο συμφέρον και τι είναι το καθήκον το οποίο <clears throat> μπορεί να φέρει πέρα σαν ένα μέλο σε σχέση με αυτό το δημόσιο συμφέρον. Ένα παράδειγμα Το έχω συμπεριλάβει στην περίληψή μου και θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί με τα διαβατήρια που εκδίδουν τα κράτη-μέλη. Ποιο είναι το καθήκον εδώ που μπορεί να αναλάβει ένα μέλος σε σχέση με την έκδοση διαβατηρίων. Μπορεί κανείς να, να ορίσει ευρύτατα καθήκοντα εδώ, δηλαδή την έκδοση διαβατηρίων σε σχέση με την κατάρτιση μετροπολιτών. Αλλά για τη συλλογή αυτών των δεδομένων, ποια δεδομένα θα συλλέγονται, πόσο καιρό θα αποθηκεύονται, πώ θα μεταφέρονται στι αρμόδιε αρχέ, θα έχουν πρόσβαση τρίτα μέρη. Ε, η πρόσβαση των τρίτων μερών, δηλαδή στα εθνικά μητρώα κατοίκων λόγου χάρη, είναι ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να αποσαφηνίζεται. Είναι κάτι που θα πρέπει να αποσαφινιστεί στην όλη νομοθετική διαδικασία. Κατά την άποψή μου, ακόμη το περιθώριο λιγμών των κρατών μελών προ αυτό δεν είναι ε, ξεκαθαρισμένο. Έπειτα, το ένομο συμφέρον που θα μπορεί να ασκεί ο ελεγκτής, το άρθρο 6 σιγματά. Εδώ, το ένομο συμφέρον σε περίπτωση που ένας ιδιώτης δώσει το δικαίωμα στον ελεγκτή να επεξεργαστεί τα δεδομένα του. Πώς ε, θα θεωρούνται ένομα τα καθήκοντα των ε, ελεγκτών, ιδιωτών, εφόσον ε, ισχύει το άρθρο 6 σήματα, διότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πέφτει σε αχρηστία. Θα πρέπει να υπάρχει ενδεχομένω μια σύμβαση, όπως λέει το άρθρο 6β. Αλλά η σύμβαση δεν μπορεί να ε, αναστέλλεται αν υπάρχει ένομο ιδιωτικό συμφέρον. Θα πρέπει το κρατικό συμφέρον να υπερισχύει και να διέπει τη σύμβαση αυτή. Αυτέ και πολλέ άλλε διευκρινήσει νομίζω θα πρέπει να μα κάνουν να μελετήσουμε ξανά και ξανά τα σημεία αυτά και να συμπεριλαμβάνονται στο κανονισμό. Θα επανέλθω λοιπόν στην ε, πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι ακόμη ασαφή. Είναι πολύ ε, είναι ευρύτατα και θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Με την ισχύουσα πρόταση θα έχει βρει πεδίο αρμοδοτήτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά γύρονται ανησυχίε σε σχέση με τον πρωτογενή νόμο. Διότι τα ουσιαστικά, τα ουσιώδη σημεία του θα πρέπει να μπορούν να γίνονται σεβαστά, κάτι που δεν επιτρέπει η τωρινή πρόταση. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε από τώρα πολύ προσεκτικά τι συνέπειε. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. Also... Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που τήρησατε το χρόνο σας. Τώρα δίνω το λόγο στους, στον επόμενο ομιλητή, τον ε, Ζων Γκονιέ. Το ίδιο λάθος κάνω πάντα. Γκονιέ, διευθυντή πολιτικής προστασίας του ιδιωτικού βίου για την ε, Microsoft Ευρώπης. Ήσασταν όμω προηγουμένω και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, άρα μπορείτε να δώσετε διαφορετικέ εναλλακτικέ. Ε, και... Ευχαριστώ. Δράττουμε τις ευκαιρίες για να εκφραστώ στη μητρική μου γλώσσα. Δεν θα μιλάω γρήγο Να αναφερθώ σε κάποια σημεία. Ευχαριστώ τον κύριο Σιγητή. Καλημέρα σε όλους σας. Παρόλο που μιλάω στα γαλλικά, θα υπάρχουν πολλές εκφράσεις, λέξεις ε, αγγλικές. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω, να επιμένω μάλλον, όταν βλέπω του, του τίτλο εδώ της ε, συνεδρίασεων στα, στη συνεδρίαση για τη μεταρρύθμιση του, του πλαισίου πλαστασίας. Θα ήθελα να σου πω ότι αυτό που είναι βασικό είναι να δημιουργήσουμε προστασία πρέπει να δημιουργήσουμε προστασία και ειδικά όταν μιλάμε για cloud computing, δηλαδή το λεγόμενο νέφος, ε, θα μπορούμε να προβλέψουμε τις εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Όταν χρησιμοποιείτε το Twitter ή το Facebook με τέτοια συχνότητα που όμως πριν από τρία χρόνια ακόμα κανείς δεν χρησιμοποιούσε, καταλαβαίνετε πόσο ραγδαίες είναι οι εξέλιξη Άρα χρειάζεται ένα πλαίσιο, ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης για τα επόμενα 20 χρόνια ενδεχομένω τελευταία νομοθεσία ήταν πριν από 17 χρόνια, νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε ότι μια ρύθμιση θα ισχύει στα επόμενα 20 χρόνια. Εγώ όταν είχα την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, την πανεπιστημιακή σταδιοδρομία στην οποία αναφερθήκατε το 2001, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια έκτοτε, ε, και γι' αυτό ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να μιλήσω ενώπιον σα για το θέμα αυτό. Τρία-τέσσερα θέματα μόνο θα ε, εκθέσω μέσα στα 10 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου, σας διαβεβαιώ. Μια επιχείρηση λοιπόν, μια επιχείρηση είτε είναι αυτή η Microsoft είτε η αδίποτε μικρομεσαία επιχείρηση και ιδιώτης ε, ε, πρέπει να, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη να έχει καταρχάς σαφείς κανόνες. Για να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη πρέπει να υπάρχουν σαφεί κανόνε. Δεν μπορούμε να αρχίζουμε να παίζουμε και στην πραγματική ζωή χωρί να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιοι είναι οι κανόνε του παιχνιδιού. Ακριβώς εδώ λοιπόν θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο, ακριβώς εδώ θα πρέπει να επιμείνουμε στο τι χρειάζεται να αναπτυχθεί ή να περαιτέρω στο κείμενο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Καταρχά, χρειάζεται μια πραγματική εναρμόνιση. Όλε οι επιχειρήσει με τι οποίε έχετε επικοινωνήσει και φαντάζομαι όχι μόνο αυτέ, ε, μεγάλοι υποστηρικτέ, φαν θα λέγαμε, του ε, της να έχει μια κατά το μέγιστο αρμόνιση να προτείνει το κείμενο αυτό και να είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, κανονισμός. Τι σημαίνει μέγιστη εναρμόνιση. Εμεί έχουμε διάφορε ιδέε να προτείνουμε. Εναρμόνιση για μα. σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφή συνένεση ως προς την ε, ε, ιδέα του κύριου ε, της κύριας έδρας. Ε, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μια επιχείρηση θα, θα έχει ε, να, της μονοθυριδικής μάλλον προσέγγισης θα έχει μια επιχείρηση να ασχοληθεί μόνο με μία αρχή να μην αναζητεί δηλαδή διάφορες αρχές με τις οποίες θα επικοινωνεί θα πρέπει ενδεχομένω βεβαίω να υπάρχει μια πρωτογενή ή δευτεροβάθμια ή δεν ξέρω τι αρχή, αλλά πάντω θα πρέπει να είναι σαφή η εικόνα για τι επιχειρήσει, μια βασική αρχή επικοινωνία. Δεύτερο παράδειγμα. Εμεί, Microsoft. Που είμαστε και επεξεργαστέ, προσέσω, αλλά και ελεγκτέ, και εδώ είναι πολύ σημαντική η όρη, ίσω ε, δεν ε, του ε, συζητούμε αρκετά συχνά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό όταν μια εταιρεία είναι και, έχει και τι δύο δραστηριότητε να, υφίσταται, να υπάγεται μόνο σε μία κύρια, σε ένα κύριο φορέα. Ε, δεν μπορεί δηλαδή τη Δευτέρα με τη μία ιδιότητα να απευθύνομαι σε ένα φορέα, φορέα και την Τρίτη σε έναν άλλον, γιατί ουσιαστικά τι ζητάμε, να ε, ασφάλεια δικαίου, προβλεψιμότητα, σαφήνεια στις διατάξεις. Όταν λοιπόν μια επιχείρηση έχει και δραστηριότητες επεξεργασίας αλλά και δραστηριότητες ελέγχου, δεν έχει σαφή εικόνα απέναντί της. Επίσης, το τρίτο σημείο, σαφής ορισμός για το τι σημαίνει επεξεργαστής και τι σημαίνει ελεγκτής για να είναι σαφής ε, η πορεία στην οποία έχουμε αποδειθεί και με ενδιαφέρον βλέπω ένα έγγραφο εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άρα στον κατάλληλο χώρο το συζητούμε πριν από μερικές ημέρες εκδόθηκε από την Γενική Διευθύνση της Ιστορικής Πολιτικής ένα έγγραφο λοιπόν με ένα πολύ χρήσιμο καταρχάς το έγγραφο είναι πολύ καλό θα σας καλέσω να το διαβάσετε όλοι ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο ως προς το τι μπορεί να βελτιωθεί στο σχέδιο κανονισμού όπου αναφέρεται ξεκάθαρα ότι τα προτινόμενα αυτή τη στιγμή με το νέο ορισμό για τον data controller, δηλαδή να ασχολείται να ε, ελέγχει το purpose, condition and means, δηλαδή το στόχο, του όρους και τα μέσα, δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στο, σε δεδομένα του cloud, γιατί δεν μπορεί ένας ελεγκτής να επαληθεύσει το condition και means, τα μέσα και τις συνθήκες. Αυτό λοιπόν που προτείνεται στο έγγραφο του Κοινοβουλίου είναι ο ρόλος του ελεγκτή ε, των δεδομένων να, είναι να επαληθεύει μόνο ε, το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, το purpose δηλαδή μόνο. Και αυτό είναι το μόνο δυνατόν που μπορεί να γίνει. Σε αυτό επιμένουμε ιδιαίτερω. Τώρα, στα τελευταία πέντε λεπτά που μένουν, θα ήθελα να επαναλάβω ότι πρέπει να είναι σαφεί οι κανόνε, ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσφυγή σε ένα μόνο φορέα και να είναι σαφή η εικόνα με ιδιαίτερη υπογράμμιση στη μελέτη αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι πολύ σωστή και εύστοχη. Στη συνέχεια. για να υπάρχει εμπιστοσύνη. Πρέπει να ξέρουμε ουσιαστικά υπό ποιου όρου παίζεται το παιχνίδι, με ποιε προποθέσει και ποιε κυρώσει σε περίπτωση που κάποιο παραβεί του όρου ε, του παιχνιδιού. Άρα λοιπόν, και εδώ αναφέρομαι στο άρθρο 79 με τις διοικητικές κυρώσεις, κύρωση επιβάλλεται Εάν κάποιος εσκεμμένα δόλια προκαλέσει ζημία, cause harm, πολύ καλά, σωστό είναι. Προφανές είναι ότι όταν κάποιο δεν τηρεί τους κανόνες του ιδιωτικού βίου να τιμωρείται, πολύ καλά και αυτονόητο. Αλλά ταυτόχρονα και για αμέλεια μπορεί κανείς να ε, υποστεί και μάλιστα μέσα στην ίδια διάταξη, στο ίδιο άρθρο μέσα. Ε, αλλά εδώ θα έλεγα προσοχή. Πώς, τι σημαίνει επιβάλλω κυρώσει σε μια επιχείρηση για ε, παραβίαση λόγω αμελίας. Εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορεί κανείς μόνο για αμέλεια να τιμωρηθεί. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχει παραβεί το καθήκον επιμέλειας προηγουμένως. Ε, ή τα υπόλοιπα καθήκοντα. Και κυρία Καραμανλή, μιλήσαμε για κατεξουσιοδότηση πράξης. Δεν θα κάνω σχόλιο προς την τοποθέτηση αλλά για τις κατεξουσιοδότηση πράξης θα έλεγα ότι καλό είναι να μην συνδεθούν αυτή τη στιγμή με την επιβολή, σε αυτό το χρονικό σημείο τουλάχιστον, με την επιβολή χρηματικού προστήμου. Ε, το πρόστιμο έχει σαν χαρακτηριστικό ότι είναι ευέλικτο μέσον και εξελίσσεται και το ίδιο το χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται μέσω εξουσιοδότηση πράξη. Αυτή τη στιγμή όμω δεν είναι σαφέ το τι είδου πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται. Αυτό θα συνδεθεί με κάποιου τεχνικού κανόνε, με κάποιε προποθέσει που ακόμη δεν είναι γνωστέ και έτσι η επιχείρηση δεν μπορεί να τιμωρείται με κάτι το οποίο είναι άγνωστο και το οποίο υπάγεται σε έναν χωριστό, σε ένα χωριστό σύνολο κανόνων. Χρειάζεται προβλεψιμότητα, το επαναλαμβάνω, και μην, σκέφτεστε ότι σα μιλάει η Microsoft. Σκεφτείτε μια μικρομεσαία ευρωπαϊκή επιχείρηση με 250 εργαζομένους το πολύ που πρέπει να γνωρίζει τι θα την περιμένουν τα επόμενα 3-4 χρόνια και τα δύο χρόνια ακόμα είναι πολύ και στα δύο-τρία λεπτά που μου μένουν θα ήθελα να πω τα εξή, ότι υπάρχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό προ την εμπιστοσύνη, τη δημιουργία του αισθήματος εμπιστοσύνη, ότι δηλαδή πρέπει να εξασφαλίσετε η δυνατότητα, πρέπει να προσφέρετε πεδίο για ανάληψη πρωτοβουλία από τον ε, επιχειρηματή, από την επιχείρηση, να υπάρχουν κίνητρα δηλαδή, ώστε να συμπεριφέρεται σωστά η επιχείρηση, ενδεχομένω με το κίνητρο της πιστοποίηση, του certification, με ένα κώδικα συμπεριφορά που μπορεί να προσδώσει πραγματική ε, δύναμη, ε, ένας κώδικας συμπεριφοράς που επιβάλλεται σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, πάντως η γενική φιλοσοφία του κειμένου είναι η εξή ότι δίνονται πολλά δικαιώματα στους data subject, δηλαδή στους στα υποκείμενα, όλους τους δικαιούχους δηλαδή, που είμαστε όλοι εμείς, το δικαίωμα στην προσφυγή και τα λοιπά, right of complaint, πολύ καλά, αλλά πρέπει και η επιχείρηση να έχει όχι μόνο υποχρέωση, να έχει και εκείνη επιπλέον δικαιώματα τα οποία πρέπει τώρα να διευκρινιστούν το Code of Conduct, το Certification, ο κώδικα συμπεριφορά δηλαδή και η πιστοποίηση, πρέπει μέσα από νέε διαδικασίε να εξελιχθούν για να διευκολύνουν τι επιχειρήσει. Και για να κλείσω στα δύο λεπτά που μου μένουν, θα ήθελα να φερθώ σε ένα ουσιοδέστατο σημείο που, αφορά, που συμπορεύεται με την έννοια τη εμπιστοσύνη και που θα πρέπει νομίζω να χαρακτηρίσει τη γενική φιλοσοφία του κειμένου, έστω και αν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμη. Εμπιστοσύνη χωρί διαφάνεια δεν μπορεί να υπάρχει υπάρξει trust ίσον transparency, εμπιστοσύνη ίσον διαφάνεια και ξέρω ότι μερικές φορές ε, μπορεί να μην καταγράφεται ρητά με στο κείμενο η διαφάνεια, αλλά αποδεικνύεται, όπως και η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη δεν ε, εντέλεται, γιατί την εμπιστοσύνη την κερδίζει κανείς και την αποδεικνύει. Το ίδιο και η διαφάνεια. Πρέπει να υπάρχουν κείμενα, παραδείγματι, που χρεώνουν το φορέα να είναι διαφανή. Στο άρθρο 29 του Position ε, Paper, παραδείγμα του προηγούμενου Ιουλίου, που υπήρχε η έννοια της διαφάνειας και πολλές προτάσεις που γίνονται εκεί πέρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Διαφάνεια για το cloud, παραδείγματι, υπάρχει ένα σύννεφο, ένα νέφος, για το οποίο γνωρίζουμε μέσα σε αυτό τι υπάρχει και αυτό πρέπει να καταστεί σαφέ, πρέπει να καταστεί διαφανέ, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια χωρί ε, ιδιωτικό βίο, δεν μπορεί να υπάρχει ιδιωτικό βίο χωρί διαφάνεια και είναι υποχρέωση τη κάθε επιχείρηση να, έχει, να εξασφαλίσει του όρου διαφάνεια. Εσεί ω πολίτη θα πρέπει, ε, παραδείγματι, έχετε το δικαίωμά σα να βάλετε στην πόρτα σα τον Do Not Disturb, μην ενοχλείτε. Ε, το ίδιο και η επιχείρηση θα κάνει ε, την προσπάθειά της για τη διαφάνεια. Δεν θα σας εκθέσω τώρα τι έχει κάνει η Microsoft που έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για τη διαφάνεια. Αλλά πάντως νομίζω ότι και οι κανόνες της συνύπαρξης, της συμβίωσης επιβάλλουν να είναι σαφείς και διαφανείς οι συνθήκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκονιέ. Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Ροντριγκέ. η οποία είναι προϊστάμενη της BOIC, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταναλωτών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον Καταναλωτών, και σας καλωσορίζω, σας δίνω το λόγο για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή ΛΥΠΕ για τη σημερινή πρόκληση. Εμείς, ε, η Μπούικ, ε, εκπροσωπούμε 42 εθνικές ενώσεις. Μπορεί να μην μας γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, εδώ είναι η έδρα μας, και ακριβώς ε, συνενώνονται σε εμάς οι εκπρόσωποι 42 ανεξάρτητων και αξιόπιστων εθνικών ενώσεων καταναλωτών. Θα ήθελα εδώ να σας παρουσιάσω τις δικές μας σκέψεις για το πώς βλέπουμε αυτήν την πρόσφατη πρόταση για κανονισμό για την προστασία δεδομένων και μετά ίσως περάσω και σε κάποιες λεπτομέρειες για τα δικαιώματα προστασίας. Εάν έχω αρκετό χρόνο θα ήθελα να σχολιάσω και τις ε, νομικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων. Γενικές λοιπόν παρατηρήσεις για το σχέδιο κανονισμού. Η η Ένωση των Καταναλωτών μας καλωσορίζει τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Πιστεύουμε ότι σε γενικές γραμμές το σχέδιο κανονισμού αποτελεί μια σημαντική βελτίωση. Υπόθηκε ήδη αρκετέ φορέ σήμερα το πρωί. Αποτελεί βήμα προόδου σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση και για την προστασία των δεδομένων και για τους καταναλωτές. Πιστεύουμε επίσης ότι η πρόταση εξευρίσκει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ από τη μια της ανάγκης για ένα πραγματικό αποτελεσματικό σύστημα προστασίας δεδομένων και από την άλλη οι επιχειρήσεις να μην πρέπει να αντιμετωπίζουν ε, υπερβάλλον διοικητικό Οι προκλήσεις ε, μπορεί να προκύπτουν και από τα πολλαπλά επιχειρηματικά μοντέλα που πλέον διαχειρίζονται και εξαρτώνται από τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Υπ' αυτό το φως το μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει το δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο. Και αυτό να μην υπονομεύεται, γιατί μπορεί να είναι πιο επικερδές να παραβιάζεται ιδίως στον εικονικό ψηφιακό κόσμο. Η βασική μας ανησυχία υπόθηκε από τον κύριο Γκονιά της Microsoft και χαίρομαι που άκουσα ότι και για εσάς είναι πολύ σημαντική η διαφάνεια. Βασική μας λοιπόν μέρημνα, ε, ανησυχία μάλλον, είναι η έλλειψη διαφανούς πληροφόρησης και ενημέρωσης από τις επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές. Ισχύει για κάποιες επιχειρήσεις περισσότερο από ό,τι για άλλες. Πολύ συχνά οι καταναλωτέ δεν γνωρίζουν ότι συλλέγονται τα προσωπικά του δεδομένα, ότι την χάνουν επεξεργασία και κάποιε φορέ είναι κατοικείμενο εμπορία πλέπει προς να το ανέχονται. Αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Δεν είναι μυστικό ότι οι σημειώσεις περί ιδιωτικής προστασίας είναι δύσκολο και να παρουσιαστούν και να κατανοηθούν από το μέσο καταναλωτή. Τι κάνουν συνήθως οι καταναλωτές αντί να διαβάζουν τις λεπτομέρειες, ε, ουσιαστικά ε, αναγκάζονται να εμπιστευτούν τι εξορισμού ρυθμίσεις, default ρυθμίσεις όπως λέγονται. Αλλά είναι τόσο πολύ σύνηθε ε, να μην καταλαβαίνουν ε, τις λεπτομέρειες λόγω του νομικού λεξιλογίου που χρησιμοποιείται, που γίνονται όλα αυτά πολύ δυσνόητα και δύσχριστα. Πέραν αυτών, όπως είπα και από την αρχή, η νέα πρόταση ε, περιέχει τα κύρια στοιχεία και ευχαριστούμε για αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διασφαλίζουν στους καταναλωτές καλύτερη ενημέρωση για το πώ χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που τους αφορούν. Και Επίση, σε ένα βαθμό αποκαθίσταται και ο έλεγχο των ίδιων των καταναλωτών στα προσωπικά του δεδομένα. Η πρόταση θα βελτιώσει την κατάσταση των καταναλωτών όποτε υπάρχει παραβίαση τη προστασία δεδομένων με ενημέρωση, χρέωση ενημέρωση για την παραβίαση των δεδομένων οριζοντίω, όχι μόνο για του ελεγκτέ ή για τι ενώσει. Από την άλλη, η πρόταση καθορίζει και το δικαίωμα των ενώσεων ή των πολιτών, των ατόμων δηλαδή, να προσφύγουν και στη δικαιοσύνη σε περίπτωση παραβίασης της προστασίας. Θα περάσω τώρα σε κάποιες λεπτομέρειες προς το τέλος της παρουσίασής μου για την επιβολή των ε, μέτρων, των νόμων μας. Τώρα, για τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους πολίτες. Η Ένωσή μας καλωσορίζει τη συμπερίληψη της νέας αρχής της διαφάνειας του άρθρου 11 και την ενδυνάμωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης, τουλάχιστον σε σύγκριση με την ισχύουσα οδηγία. Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα λήθης ή διαγραφής όπως ονομάστηκε, μπορούμε να στηρίξουμε, μπορούμε να συμφωνήσουμε με, την νέα, με το νέο αυτό στοιχείο, ώστε να ενδυναμώνεται το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων. Πολλές φορές στο επιγραμμικό περιβάλλον ε, το δικαίωμα αυτό της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων παραμγωνίζεται πλήρως. Θεωρούμε όμως ότι η έννοια της λύθης μπορεί να είναι παραπλανητική για τους καταναλωτές. Το είπα και προηγουμένως εδώ πριν από λίγα λεπτά. Στην πράξη υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στι δυνατότητε διαγραφή σβησίματο των προσωπικών δεδομένων στο ψηφιακό περιβάλλον. Πρώτον, το δικαίωμα στη λύθη σε μερικέ περιπτώσει μπορεί να μην είναι συμβατό με την αρχή τη ελευθερία του λόγου, Επιπλέον, η υλοποίηση του δικαιώματο αυτού στη λύθη, στη διαγραφή και η η επιβολή του, η υλοποίησή του, μπορεί να μην συνάδει με τα τεχνικά μέτρα που προκύπτουν από τα φίλτρα των ψηφιακών ε, μέσων επικοινωνίας. Έπειτα όλα τα τρίτα μέρη στα οποία έχουν αποκαλυφθεί τα δεδομένα μπορεί να μην ε, ασκήσουν με τον ίδιο τρόπο το δικαίωμα αυτό διαγραφής. Είναι λοιπόν μια υποχρέωση που έχει να κάνει με την προσπάθεια, αλλά δεν θα υπάρχει αναγκαστικά το επιδιωκόμενο τελικό αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρξει απαραίτητη νομική βεβαιότητα για αυτό την αρχή. Είναι καθοριστική σημασία η λύθη, εφόσον μιλάμε για προστασία δεδομένων και τον εξασφαλιστή. Η φορητότητα τώρα, η δυνατότητα μεταφορά των δεδομένων, αυτό είναι ένα νέο δικαίωμα το οποίο δεν υπάρχει στην ισχύουσα νομοθεσία. Αλλά δεδομένων των εξελίξεων στις τεχνολογίες της επικοινωνίας, ε, καλωσορίζουμε πραγματικά την ε, πρόβλεψή του. Έχουμε λάβει εκθέσεις από τα μέλη μας που δείχνουν ότι σήμερα όταν οι καταναλωτές αποθηκεύουν πληροφορίες σε συγκεκριμένες πλατφόρμες ή υπηρεσίες όπως τα κοινωνικά δίκτυα ή στα email τους, Πολλέ φορέ δεν μπορούν να μεταφέρουν τα δεδομένα αυτά από τον ένα παροχέα υπηρεσιών στον άλλο. Οι περισσότεροι διεκδικούν την αποκλειστικότητα της αποθήκευσης των δεδομένων στα δικά τους αρχεία. Η κατάσταση αυτή προφανώς δεν είναι συμβατή με τα δικαιώματα των καταναλωτών να ελέγχουν οι ίδιοι τα δεδομένα τους και ε, να μπορέσουν να αρνηθούν την επεξεργασία των δεδομένων τους. Επίσης εμποδίζεται ο ανταγωνισμός μεταξύ της ε, μεταξύ των παροχών, παροχιών υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται δηλαδή η μετάβαση από τον ένα παροχή στον άλλο. Ε, η συμπερίληψη τώρα της κατάρτισης, ε, μέτρων για την κατάρτιση προφίλ στο σχέδιο κανονισμού. Είναι κάτι που επίσης καλωσορίζουμε. Στην ισχύωση οδηγία υπάρχει ως έννοια, αλλά εδώ διευκρινίζεται καλύτερα τα μοντέλα διαφήμισης των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται τα προφίλ των πολιτών και των ατόμων στο διαδίκτυο είναι πολλαπλά. Όμως οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τις πρακτικές αυτές διαφήμισης. Τους ανησυχούν, αλλά δεν τα γνωρίζουν. Δεν ξέρουν ακριβώς με τι έχουν να κάνουν. Δεν γνωρίζουν ούτε τα μειονεκτήματα, ούτε τα πλεονεκτήματα, ούτε τις ε, ε, επιπτώσεις της κατάρτισης προφίλ. Συνολικά, στηρίζουμε τη γενική προσέγγιση του σχεδίου κανονισμού σε ό,τι αφορά την κατάρτιση προφίλ, όμω χρειάζονται προσθήκε στα μέτρα αυτά, ώστε οι καταναλωτέ να μπορούν οι ίδιοι να ελέγχουν τα δεδομένα του. Πρώτα απ' όλα, το δικαίωμα να αρνηθούν την κατάρτιση προφίλ θα πρέπει να συνοδεύεται αυτό με το δικαίωμα ενημέρωση, με τρόπο φιλικό μάλιστα για τον καταναλωτή. Να γνωρίζουν τι τεχνικέ και τα μέτρα που χρησιμοποιούνται από το οικοσύστημα τη διαφήμιση, αλλά και για τι σημαντικέ επιπτώσει που μπορεί να έχουν τα μέτρα αυτά στου ίδιου εφόσον για αυτούς λέγονται τα δεδομένα. Έπειτα, στηρίζουμε την ε, υποχρέωση ενημέρωσης για παραβίαση προστασίας δεδομένων, διότι μπορεί να βλάπτονται οι καταναλωτές, μπορεί να βλάπτονται οι καταναλωτές από την ε, άσκοπη αποκάλυψη των τραπεζικών τους λόγου χάρη στοιχείων, ε, αλλά το ίδιο και από το, την αποκάλυψη των στοιχείων των τηλεφωνικών τους ε, λογαριασμών λόγου χάρη. Είναι πολύ καλή λοιπόν αυτή η υποχρέωση ενημέρωσης για την παραβίαση δικαιωμάτων. Ε, σε κάθε περίπτωση είναι αρνητικές οι συνέπειες για τους πολίτες και θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση εφόσον υπάρχει παραβίαση, ώστε να μην υπάρχει αλλά μόνο σε περίπτωση που είναι σημαντικές οι παραβιάσει ώστε να μην επέλθει και η λεγόμενη κόποση των, ε, της ενημέρωσης, της πληροφόρησης. Θα πρέπει επιπλέον το κόστος της βλάβης να είναι αντικείμενο αποζημίωσης, προκειμένου να, είναι, να έχει νόημα αυτή η υποχρέωση. Θα πρέπει να προβλεφθεί και σε δικαστικό επίπεδο η επιβολή αυτή αποζημιώσεων. Θα πρέπει να μπορεί ο πολίτης, το άτομο ή ενώσεις καταναλωτών, ομάδες καταναλωτών να μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Συλλογικές λοιπόν προσφυγές ε, σε περίπτωση που θέλουμε να υπάρχει πραγματική υποχρέωση ενημέρωσης. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει το χρόνο μου. Οπότε να επαναλάβω ότι καλωσορίζω την ε, πρόταση αυτή και θα περιμένω και τις ερωτήσεις σας. Με χαρά θα τις απαντήσω στη συνέχεια της, ε, του διαλόγου μας. Σας ευχαριστώ. Thank you also. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και... Κύριος Ντέινς, καθηγητής από το London School of Economics, γνωστός για την έρευνά του στον, στην προσφυγή του ιδιωτικού βίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω σήμερα. Θα είμαι όσο δυνατόν πιο σύντομος, αναγκαστικά, για να δώσω τη σύντομη ιστορία Πριν από το καλοκαίρι οι συντάκτες εκθέσεως ε, για τα θέματα αυτά μου ζήτησαν να κάνω μία μελέτη της, ε, της μια αξιολόγηση των εμπλεκομένων ε, και των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων. Πρέπει να πω ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα από μένα αυτά. Η βασική ιδέα ήταν μία βασική Ήταν μια βασική αξιολόγηση της ε, μακροπρόθεσμης δομής. Αυτό χρειάστηκε να κάνουμε λοιπόν και θα σας δώσω πρώτα την καλή είδηση ότι περάσαμε το καλοκαίρι Συνομιλώντα όχι με του συνήθει υπόπτου, γιατί ξέρετε ότι το 90% των απαντήσεων το παίρνουμε από του ίδιου πάντα φορεί. Όχι, το περάσαμε μιλώντα με 2-3 χιλιάδε ιδιώτες ε, και κάποιε ε, ιστοσελίδες ε, μέσω κάποιων σελίδων κοινωνικών δικτύων αλλά και σε συνεδριάσεις. Και έτσι καταγράψαμε τις απαντήσεις τους, τις προτάσεις. Η καλή είδηση λοιπόν και αυτό θα είναι η σύντομη ε, το σύντομο κομμάτι, ότι φαίνονται οι αρχές λογικές και τα θεμέλια του κανονισμού φαίνονται φαίνεται να έχουν ε, σχετικά γενική υποστήριξη ακόμη και από τους πιο επιφυλικτικούς. Αυτή είναι η καλή είδηση λοιπόν για τα θεσμικά όργανα. Επίσης, φαίνεται ότι οι υποδομές για την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη γενικά τη χάνει υποστήριξης και θα έλεγα συντριπτικής υποστήριξης. Αυτά είναι τα καλά νέα λοιπόν. Από την άλλη, η επιπλοκή όπως θα λέγαμε ευγενικά, είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία προς ούτε καν ένα συγκεκριμένο σημείο του κανονισμού, συνένεση που να καλύπτει τους πάντες δηλαδή. Και αυτό νομίζω γιατί υπάρχουν δύο παρακαταθήκες. Πρώτον, από την οδηγία του 1995 υπάρχει μια σημαντική και εκτεταμένη αντίληψη και ευαισθητοποίηση ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το 85% των συζητήσεων είχε να κάνει με τον ιδιωτικό τομέα. Το 80% των συνομιλιών που κάναμε εμείς στη διαβούλευση του ε, London School of Economics είχε να κάνει με το δημόσιο τομέα και ανησυχίε για έναν μεγάλο αδελφό Big Brother έλεγχος και εποπτεία είναι βασική ανησυχία του κοινού, όπως άλλωστε καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι η πρώτη επιπλοκή. Το να πείσουμε το κοινό δηλαδή για τις επιλογές. Και πάλι, για να μιλήσω ακόμη για το γενικό κοινό, δεύτερη παρατήρηση, η αίσθηση ότι έχουν αποτύχει θεσμικά οι αρχές οι αρμόδιες για τη ρύθμιση προστασίας των δεδομένων. Δεν υπάρχει ενιαία νομοθεσία, δεν υπάρχει εφαρμογή, δεν υπάρχει αντίληψη όμως παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποτυχία αυτή. Στη Γερμανία, Φερρυπίνη, στις χώρες δεν αισθάνονται ότι έχει αποτύχει όπως το κοινό το οποίο είδαμε εμείς. Στην υπόλοιπη Ευρώπη όμω η έννοια αυτή τη αποτυχία, η ιδέα ότι έχουν αποτύχει τα ευρωπαϊκά όργανα, όχι εθνικέ αρχέ απαραίτητα, αλλά εν γέννη και συλλήβη ότι έχει αποτύχει το κράτο δικαίου, φτάνει μέχρι την κοινική αντιμετώπιση και θεώρηση κατάστασης. Άρα, από το 1995 μέχρι τώρα έχουμε αυτές τις δύο παρακαταθήκες, κοινωνικές, πολιτιστικές γραμμές που καθοδηγούν την αντίληψη του κοινού και ως εκ τούτου την υποστήριξη των εμπλεκομένων φορέων ή την αντίθεσή τους στις προτάσεις. Όταν άρχισαν λοιπόν, άρχισα να ανάγομαι στο χρόνο αυτής της πρότασης και να την ε, αποκαλύπτω φίλο-φίλο μέχρι τον πυρήνα της, είδα ότι υπάρχουν διάφορες ε, θέσεις από τους εμπλεκομένους φορείς ανά τα έτη που έχουν εκφραστεί. Αλλά θα ήθελα ιδιαίτερως να επισημάνω προς μηχανισμούς μία ιδέα που φαίνεται να επικρατεί σαν να υπάρχει κάποιος, κάποιο οικουμενικό δίκαιο, οικουμενικός νόμος, σαν τους νόμους της φυσικής, που ισχύουν πάντα, ό,τι δηλαδή. Όταν καλείται ένας ε, φορέας να προβεί σε ορισμούς, να περιγράψει δικαιώματα ή κύκλους συμφερόντων ή να δώσει ένα επακριβή ορισμό ενός τομέα θεσμικά, τότε η, ο κλάδος ο οικονομικός, οι επιχειρήσεις δηλαδή, έχουν την αντίστροφη ή την αντίθετη τάση. Το ίδιο και αντίστροφα. Οπότε επιδιώκει κάτι ο επιχειρηματικό κόσμος, οι πολίτες θέλουν ακριβώς το αντίθετο. Δεν μπορώ να καταλήξω συμπεράσματα, δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα από αυτό το φαινόμενο, αλλά το καταγράφω. Θα υποβάλω τα έγγραφά μου βέβαια στη γραμματεία τόσο λίγο για να προβώ τι ε, περιγραφές και τα, τα, την εικόνα που μας δίνουν οι ιδιωτικές αυτές έρευνες που έχουμε κάνει. Αλλά πάντως καταλήγω στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να, να προσπαθήσουμε να φέρουμε πιο κοντά τα δύο αυτά άκρα, να εξορροπήσουμε αυτή την ε, εξίσωση, ούτω ΣΥΚΠΗΝ, ώστε να έρθουν πιο κοντά τα δύο άκρα, πράγμα το οποίο όμω δεν θα είναι εύκολο γιατί θα πρέπει να διαγνώσουμε ποια είναι η δυναμική του προβλήματος πρώτα απ' όλα. Και υπάρχουν 28 θέματα βασικά θέματα που εμφανίζονται διαρκώς στην, ε, στον κανονισμό για τα οποία όλοι συμφωνούν ότι χρειάζονται περισσότερο αυστηρούς ε, ορισμούς και περισσότερη διαφάνεια. Στην ε, κορυφή αυτής της λίστας, αυτού του καταλόγου, είναι από την πλευρά του κοινού ο ρόλος των Εθνικών Αρχών Δεδομένων όχι μόνο ως προς τις εξουσίες της αρχής αυτής, αλλά και ως προς την αιμονή της στην εκτέλεση του έργου του, της tenacity στα αγγλικά. Αυτό είναι ένας όρος ο οποίος επανέρχεται παγίως στις απαντήσεις. εμονή λοιπόν και πείσμα στην εκτέλεση του έργου και τεχνικές δεξιότητες, ικανότητες. Αυτό είναι χαρακτηριστικό στις απαντήσεις που σαν σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι το εφαρμοστέο δίκαιο είναι ο δράκος που παραφυλάει μέσα στην σπηλιά του για όλους μας. Επίσης η μεταφορά σε εθνικό επίπεδο και η συνεπής εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Αλλά για να περάσω και στην μικρό μικρο λεπτομέρεια, όταν ο εμπλεκόμενος, οι εμπλεκόμενοι φορείς, stakeholders συζητούν διάφορα θέματα λεπτομερή, όπως φερειπίν ε, την προστασία του ιδιωτικού βίου, προκύπτουν ζητήματα από την εποχή παραδείγματι της τεχνολογίας ενίσχυσης της, ε, του ιδιωτικού βίου, που είναι αρχαία ιστορία για πολλούς από εμάς όσους τα γνωρίζουν δηλαδή. Και αρχίζει πάλι ο κόσμος να ε, εκφράζει ανησυχίες. Προκύπτει λοιπόν ένα απλό μήνυμα από όλα αυτά που ενισχύσαν με τις παρεμβάσεις αρκετοί από τους ομιλητές της έδρας εδώ, ότι δηλαδή η κατεξουσιοδότηση πράξης έχουν δυναμικό τέτοιο, το οποίο γεννά πολλές ανησυχίες και δυσπιστία Λίγη είναι η εμπιστοσύνη που μπορεί να εκφράσει ο πολίτης ως προς την ε, υποχρέωση λογοδοσία, την ισονομία, την δικαιοσύνη που μπορούν να φέρουν αυτές οι κατευθυντικές πράξεις και ζητεί ο πολίτης να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, δηλαδή βλέπει ότι μπορούν να γίνουν για την ε, ανάπτυξη δευτερογενών μηχανισμών οι οποίοι θα προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις, ασφάλεια δηλαδή, λειτουργίας πέραν αυτών των πράξεων καταξουσιοδότηση, ώστε να αποδεικνύεται στον πολίτη ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στο τελικό αποτέλεσμα. Από τις εκατοντάδες παρατηρήσεις που έχω εγώ σημειώσει από τη διαδικασία αυτή της διαβούλευσης, η οποία θα συνεχιστεί επαναλαμβάνω, επισημένο μάλλον και στο φθινόπωρο, τρέχον φθινόπωρο, θα πρέπει να επισημάνω ότι απολύτως κρίσιμη σημασία για την επιτυχία αυτού του κανονισμού είναι ακριβώς η ιδέα της εμπιστοσύνης. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Πολλά ενδιαφέροντα θέματα που τώρα μπορούμε να συζητήσουμε, ακούσαμε. Έχω δύο αιτήσει για να λάβουν το λόγο από μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και άλλε δύο από Ευρωβουλευτέ. Έρχονται ακόμη οι κάρτε, τώρα έχουμε τρει. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Ράχενμπαχ από την γερμανική Bundestag. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και από δικής μας πλευράς χαιρετίζουμε την ιδέα για έναν ε, κανονισμό, την ιδέα για την εναρμόνιση. Δεδομένα τα οποία έχουν ε, ιδιαίτερη αξία οικονομικής δηλαδή αξιοποίησης πρέπει ιδιαίτερα να προστατεύονται και εδώ μιλούμε όχι μόνο για την πρώτη ύλη ούτως υπήν, αλλά για το σύνολο των δεδομένων που μπορεί να έχουν τέτοια εμπορική αξιοποιησιμότητα. Επομένως βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες θετικές ε, επισημάν, κάποιες επιτυχημένες επισημάνσεις, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο σε κάποια σημεία. Ξεκινώ λέγοντας ότι πρέπει να καταστεί σαφέ ότι ο κανονισμό δεν ισχύει μόνο στον τομέα εκείνων τη επεξεργασία των δεδομένων, αλλά και εκεί μέσα στις συμβατικέ σχέσεις θα έλεγα, όπου μπορεί να χορηγηθούν στοιχεία, προσωπικά δεδομένα δηλαδή, και να καταγραφούν για λόγους επί παραδείγματι παροχή υπηρεσιών. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει προστασία ώστε τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα να μην μπορέσουν να αποκλείσουν ε, από το πεδίο εφαρμογής και προστασίας του κανονισμού τα διμερώς προσφερόμενα, συμβατικά δηλαδή προσφερόμενα δεδομένα. Επίσης, η επεξεργασία δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών από τρίτα, σε τρίτα κράτη δεν ε, θα πρέπει να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής, θα πρέπει να καλυφθεί και αυτή επαρκώς. Τρίτη παρατήρηση, πιστεύω ότι πρέπει να καταστεί σαφές ότι για να έχει υποδειγματικό ρόλο και χαρακτήρα αυτός ο κανονισμός δεν μπορεί να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογή του τα θεσμικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με την δυνατότητα ε, ε, επιβολής νομοθεσίας μέσω κατεξουσιοδότησης πράξεων. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν πρέπει να είναι υψηλό ο αριθμό των θεμάτων που θα καλούνται με κατεξουσιοδότηση πράξη. Πρακτικά, επίση, πρακτική εφαρμογή που θα πρέπει να έχουν αυτέ οι ε, διατάξει. Εδώ ξέρουμε ότι υπάρχει μία σειρά δεσμών, επαφών, δικτύων με τα οποία μεταφέρονται τα δεδομένα ενός πελάτη της μίας επιχείρησης σε μίαν άλλη ή άλλες και υπάρχει ένας τεράστιο, μια τεράστια διακίνηση προσωπικών δεδομένων Άρα λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο θα ελέγχεται αυτή η κινητικότητα των δεδομένων πρέπει πρακτικά να επιληθεί και επίσης για μια κεντρική ε, επισήμανση κλείνοντας δεν θέλω να πω ότι τεράστια σημασία έχει ε, η θέση του παιδιού σε όλο αυτό το πλέγμα πρέπει να είναι σαφής η προστασία και πρέπει να εξασφαλίσουμε προστασία ισοδύναμη τουλάχιστον με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών προστασία χωρίς να αποκλείουμε εξορισμού το παιδί από την πρόσβαση, αλλά δεν θα πρέπει να μπορεί κάποιος ε, να συλλέγει στοιχεία προσώπων που βρίσκονται ακόμη στην ανάπτυξη, που ακόμα δεν έχουν δηλαδή ενηλικιωθεί και πάνω απ' όλα να αποθηκεύει και να επεξεργάσει τα στοιχεία αυτά. Ε, όπως είπε και η κυρία Ροντρίγκε, λοιπόν, πιστεύω ότι χρειάζεται μια σαφής ρύθμιση, χρειάζεται ρύθμιση και για, τις, για την άειλη ζημία, την ηθική λεγόμενη ζημία, την ε, δυνατότητα αποκατάστασης σφαλμάτων ε, καταγραφής προσωπικών δεδομένων και αυτής της ηθικής ζημίας ή της άλλης ζημίας και επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει στον τομέα αυτών των προσωπικών δεδομένων να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες από αυτούς που ισχύουν στη λυπή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Επομένως η επιβολή κυρώσεων είναι πάρα πολύ σημαντική για μας και θα πρέπει εξάπαντος να εισαχθεί στο κείμενο του κανονισμού έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος ο οποίος αξιοποιεί ε, προσωπικά δεδομένα ψηφιακά να έχει μια ευνοϊκότερη, περιπτώσει θα βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση από αυτόν που τα αξιοποιεί σε επιχάρτου. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Βεβαίω, ε, όποιο άλλο από του ομιλητέ θέλει μπορεί να καταθέσει τι παρεμβάσει, γραπτέ παρεμβάσει εφόσον υπάρχουν ε, ή ε, να ζητήσει το λόγο. Όλοι οι βουλευτέ είναι ευπρόσδεκτοι. Ο κύριο Κάλλη τώρα από την Πολωνική Βουλή, τη ΣΕΝ, μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ το λόγο για δεύτερη φορά σήμερα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Συμμετείχα και στο προηγούμενο γύρο συζήτησης, αλλά στα πλαίσια του Υπουργείου Εσωτερικών συμμετείχα και στην ε, σύνταξη του δικού μας νόμου για την προστασία των δεδομένων. Οπότε γνωρίζω το θέμα καλά και με ενδιαφέρει και συμμετέχω και στην Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Όρνουγκ ανέφερε μια σημαντική αρχή ότι αυτός ο, η πρόταση κανονισμού δεν συμπεριλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου. Ο κύριος Χόρνουγκ μάλιστα είπε ο κύριος Γκονιέ μάλλον, μάλλον μας είπε κάτι κάπως διαφορετικό ότι όλα τα αντικείμενα επεξεργασία θα πρέπει να ελέγχονται. Ενώ ο κύριος Ντέιβις είπε ότι θεμελιώδε ζήτημα είναι, είναι το πώ οι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αποφεληθούν από αυτόν τον κανονισμό. Εγώ έχω την εξή ερώτηση. Στο πεδίο εφαρμογή αυτού του κανονισμού που ακόμη δεν είναι σαφές και δεν είναι συγκεκριμένο, θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα συμπεριλαμβάνεται. Δεδομένα, οι εμπορικέ σχέσεις ε, μέσω του διαδικτύου θα καλύπτονται και εμπορευόμενοι που δεν έχουν καμία έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καμία εγκατάσταση. Θα μπορούσαν να έχουν την έδρα τους ή την εγκατάστασή τους σε τρίτη χώρα. Και ταυτόχρονα Άλλες χώρες δεν ε, έχουν προβλέψεις ε, σε επίπεδο ανάλογο για την προστασία με αυτό που θέλουμε εμείς να καλύψουμε με τον κανονισμό μας. Επίσης, οι πολίτες, τα άτομα για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα, κάποιες φορές βρίσκονται μεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιες φορές όχι. Μπορεί να ε, είναι προσωρινά στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι Ευρωπαίοι πολίτες αναγκαστικά. Μιλώ για μετανάστες από τρίτες χώρες. Στην ε, Πολωνία ξαφνικά έχουμε γίνει πόλος έλξης για μετανάστες ε, ξανατολών. Ε, καθημερινά έρχονται κύματα μεταναστών. Εδώ λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει και με αυτά τα δικαιώματα. Και εδώ και να θυμίσω πάλι την παρέμβαση του κυρίου Χόρνου. Η ερμηνεία των διατάξεων αυτών για τους Ευρωπαίους, για, τα για, τους Ευρωπαίους πολίτες, προκαλεί και γύρει ζητήματα. Υπάρχουν ε, πιο περίπλοκες καταστάσεις. Οι Ευρωπαίοι ηθήνοντες αναγκάζονται Ε, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο κόστος για την ε, υλοποίηση των νόμων αυτών σε σχέση με, το, με όσους βρίσκονται εκτός Ένωσης. Άρα θα υπάρχει εδώ στρέμπλος συνταγωνισμού. Ερωτώ λοιπόν, με το σχέδιο αυτού του κανονισμού έχουμε τουλάχιστον ε, σκεφτεί την πιθανότητα να υπάρξουν μηχανισμοί για την υλοποίηση αυτού του κανονισμού χωρίς να παραμείνει μια ουτοπία αυτή η υλοποίηση. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Κέρια ερωτήματα. Θα προσπαθήσουμε να τα συγκεντρώσουμε. Ο κύριος ε, Μπάτσες τώρα από, τον, από την Ισπανική Γερουσία. Η κυρία. Ε, ε, Στο κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ στην παρέμβαση του κυρίου Ντέιβις. Η υπηρεσία στην προστασία των δεδομένων στην Ισπανία δουλεύει πολύ καλά. Εγώ δεν θα ήθελα τώρα εδώ πέρα να απλοποιήσω στην ανάλυση μου την πραγματικότητα. Σε Ξέρω ότι όλες οι χώρες μέλη αντιμετωπίζουν διάφορες καταστάσεις. Εμείς στην Ισπανία αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αρμόδια υπηρεσία, υπάρχει εδώ και χρόνια και είναι αποτελεσματική, επαγγελματική, είναι μια υπηρεσία ανεξάρτητη, με ικανότητε καταστολής. Ε, ε, έχουμε πολλές αποφάσεις στα δικαστήρια μας αναγνωρίζετε, δηλαδή το έργο αυτής της αρχής. Ανησυχούμε για το κανονισμό που προβλέπεται σε κοινωτικό επίπεδο, διότι η ιδέα μας φαίνεται σε γενικές γραμμές ε, καλή, να υπάρχει μια γενική ένα γενικό σημείο αναφοράς, αυτό φαίνεται πολύ θετικό για τις επιχειρήσεις, αλλά τι γίνεται στην πρακτική. Μήπως δημιουργούνται προβλήματα για τους πολίτες. Να γίνω πιο σαφής. Θεωρούμε ότι μπορεί να δημιουργήσει μια, ένα, ένα χάσμα ανάμεσα στην υπηρεσία, την αρμόδια και στους πολίτες. Σε σχέση με μια χώρα όπου τα πράγματα έχουν λειτουργήσει πολύ καλά ανάμεσα στον πολίτη και την αρχή. Αυτή η αρχή για μια νέα προσέγγιση μπορεί να, είναι πολύ περίπλοκη. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Διότι ε, αφού το έχουμε φέρει πριν τη γνωμοδότηση μιας αρμόδιας αρχής, αν η γνωμοδότηση της αρχής είναι διαφορετική σε σχέση με την προσέγγιση του, της κρότας μέλου όπου έχουμε ένα πολίτη, τι γίνεται, πώς προχωράμε, σε ποιον μπορεί κανείς να απευθυνθεί. Μπορεί να υπάρχουν δηλαδή προβλήματα όσον αφορά τις ε, τη διοικητική διαδικασία. Όταν δηλαδή αυτό το θέμα αφορά διαφορετικές χώρες. Όταν έχουμε να κάνουμε με την κατεξιοδότηση πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδώ γίνεται σαφές για μας ότι πρέπει να υπάρχει ένα διαχωρισμός ανάμεσα στην εφαρμογή του κανονισμού στις επιχειρήσεις και αυτού που αφορά τους πολίτες. η αρχή στην οποία μπορεί να ε, απευθύνεται ο πολίτη, θα πρέπει να είναι η εθνική αρχή. Αυτό είναι πιο απλό, απλή τρόπο προσέγγισης, λειτουργήσε τα πολύ καλά. Θα πρέπει δηλαδή να προσβληθεί ένα τέτοιο διαχωρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Κύριε Ντίπλ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, προς δύο από τους ομιλητές στην έδρα. Η κυρία Καχαμονλή, εάν κατάλαβα καλά, μίλησε για την ανάγκη να περιοριστεί το λεγόμενο profiling, η εξαγωγή δηλαδή συμπερασμάτων για τα χαρακτηριστικά του ε, υποκειμένου. Τι σημαίνει profiling, εάν δώσω την ε, διεύθυνσή μου, αν δώσω έναν αριθμό λογαριασμού, ο... παραλήπτης μπορεί να να συναγάγει συμπεράσματα και να προσπαθήσει να μου κάνει διαφήμιση με τα χαρακτηριστικά αυτά, πραγματοποιήσω θα μπορούσα να αποφύγω. Το θέμα όμως είναι εάν δίνει τα δεδομένα μου σε έναν τρίτο όλη αυτή τη δυνατότητα απαγόρευσης δηλαδή της χρήσης από τρίτων ε, των δεδομένων. Αυτό εννοείται. Εννοείται ότι θα πρέπει σε κάθε προσπάθεια ε, συναγωγή συμπερασμάτων για τον πολίτη. Το profiling δηλαδή θα πρέπει να δίδεται ρητά η άδεια για τα παιδιά, το αφήνω στην άκρη και το κάλυψε ο συνάδελφο από τη γερμανική Bundestag. Για τον εκπρόσωπο της Microsoft τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα των κυρώσεων και των κινήτρων που ανέφερε. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο πώς το εννοείται αυτό συγκεκριμένα. Σήμερα ήδη μία επιχείρηση θα μπορούσε να ξεκινήσει να εφαρμόζει αυτά που εμείς ακόμα συζητούμε και δεν έχουν γίνει νομοθεσία. Αυτό ναι, αυτό θα το θεωρούσα πολύ αξιόλογο και θα το επενούσα. Εάν όμως μετά τον ορισμό, μετά την ε, ε, ε, ε έγκριση της, ε, του κανονισμού μου αρχίσει να μου εφαρμόζει τα στοιχεία του κανονισμού, γιατί θα πρέπει να την επενέσω και να της δώσω κίνητρα. Είναι σαν να μου λέτε ότι εφόσον ισχύει ο κανονισμός ότι πρέπει να σταματάμε στο κόκκινο, όποιος σταματάει στο κόκκινο θα παίρνει και ένα βραβείο. Αυτό είναι το κίνητρο που ζητάτε. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κέρκοπ. Ευχαριστώ. Για... Προς τον κύριο Ντέιβις ε, ήθελα να θέσω μια ερώτηση, γιατί μας είπε ότι εκπώνησε και μια ε, μελέτη σχετικά. Ξέρετε ότι ως εισηγητής για το Ευρωπαίο μετρό τον κατάλογο επιβατών, στοιχείων επιβατών ε, και ως εισηγητής είχα αναλάβει ιδιαίτερη δράση. Ξέρω, Γιάν, ότι εσύ έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και μα έχει απασχολήσει πολύ προστασία δεδομένων και για τι κοινέ μα συμφωνίε με τον ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν, στι προηγούμενε συζητήσει μα, Έχουμε μιλήσει για τα διάφορα κέντρα επεξεργασία δεδομένων. ένα και πολλαπλασιάζονται παγκοσμίω. Και μάλιστα χρειάζονται φοβερού πόρου για να τα καταφέρουν. Τόσο πολλοί έχουν πολλαπλασιαστεί. Ακόμη και πόρου ε, σε υδροδότηση. Αυτό το συνειδητοποίησα μόλι χθε, πρέπει να σα πω. Και ε, συνειδητοποιώ ότι η συλλογή δεδομένων όλο ένα και ε, εντείνεται το ίδιο και η συλλογή προσωπικών δεδομένων αλλά και η επεξεργασία. Οι χρήσει μάλιστα των δεδομένων για εμπορικού σκοπού και αυτέ διαρκώ πολλαπλασιάζονται. Η δικαιολογημένη χρήση των δεδομένων για να προστατευτούμε από τρομοκρατικέ ή εγκληματικέ ενέργειε, νομίζω και αυτή ε, διαρκώ αυξάνεται. Και εδώ μιλώ σε ένας ταπεινός ε, νομικός, αλλά νομίζω ότι ο μισός πληθυσμός της γης ουσιαστικά περνάει το χρόνο του στέλνοντα τα δεδομένα του στον άλλο μισό πληθυσμό τη γη που επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα και τα αποθηκεύει. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι εγώ αφελώς συμπληρώνω όλα τα έντυπα που απαιτούνται. Κάθε φορά που κάτι χρειάζομαι, κάθε φορά που κάτι αγοράζω, πρέπει να συμπληρώσω ένα έντυπο. 20 ερωτήσεις, 30 ερωτήσεις, 40 σημεία. Ε, οτιδήποτε μπορεί να με απασχολεί στη ζωή και να δώσω μια περιγραφή του ε, ποιο είμαι. Αυτό θα ισχύει στο μέλλον. Ο κύριο Ντέιβι, τι φαντάζεται. Σα ευχαριστώ. Για το γύρο αυτόν λοιπόν τώρα έχουμε τον κύριο Κέλλη, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η συντάκτης ε, της νομοδότης εκ μέρους της Επιτροπής Βιομηχανίας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήρθα μάλλον να ακούσω παρά να κηρύξω νέε ιδέε. Για την κυρία Ροντρίγκε, πάντω, μια παρατήρηση. στο δικαίωμα στη λύθη. Είπατε ότι ενδεχομένω να μην είναι συμβατό με την ελευθερία τη έκφραση. Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτό. Διότι μου φαίνεται παραδοξολογία αυτό που άκουσα. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Ευχαριστώ πολύ στο μία ερώτηση. Και άρα έχουμε χρόνο αρκετό για να ακούσουμε να απαντηθούν οι ερωτήσεις από την έντρα. Και την πρώτη ευκαιρία απάντηση θα λάβει η κυρία Μαριέτα Καραμαντλή, γιατί θα πρέπει να φύγει και νωρίτερα από τους άλλους, φαντάζομαι ότι έχει κάποιο τρένο να πάρει για το Παρίσι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Σίτη. Θα μιλήσω λιγότερο. Ε, θα μιλήσω λίγο πιο σιγά, έχω μια τάση να μιλάω γρήγορα και θα φύγω νωρίτερα διότι στην ε, Εθνοσυνέλευση έχουμε σημαντικό κείμενο ε, η συνθήκη για τη σταθερότητα για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Είναι σημαντικό λοιπόν η Γαλλία, η πλειοψηφία μάλλον, να εκφραστεί. Λοιπόν, πολλά θέματα έχουν θυχθεί. Δεν θα μπορέσω σε όλες τις ερωτήσεις να απαντήσω, αλλά θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μας οδηγούν σε μια σειρά ανησυχιών που δείχνουν να είναι κοινέ. Και εγώ είμαι εδώ επίσης για να, ε, να ε, κάνω μια ανάλυση του Κοινοβουλίου, κάτι που εκφράζει τους συναδέλφους μου και χαίρομαι που άκουσα τους συναδέλφους που έχουν εκφρασίσει για τα προσωπικά δεδομένα. Ξεκινάω από το τέλος. Κάτι ελέγχθη η κυρία Σίπελ για το λεγόμενο profiling για τον περιορισμό του. Δεν είναι θέμα θρησκευτικής προσέγγισης. Το profiling μπορεί να γίνεται επικεντρωμένο, στοχευμένο. Ε, αυτό συνδέεται με το δικαίωμα στη λύθη. Αυτό έχει να κάνει με την ε, ε, διατήρηση και διόνυση των δεδομένων. Αν έχουμε ένα στοχημένο profiling, καλύτερα φυσικά μπορεί να προστατεύσει κανείς τα προσωπικά δεδομένα. Και αναφέρουμε εδώ πέρα σε ψηφίσματα τα οποία έχουν γίνει από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μου φαίνεται όμως ότι ο διεισηγητής δείχνει την ανάλογη ευαισθησία και το έργο θα συνεχιστεί. Επίσης, να πω κάποιο άλλο στοιχείο τώρα. Ε, δόθηκε μια έμφαση στις αναλύσεις μας σε αυτό το οποίο μπορεί να βελτιωθεί. Υπήρξε πρόοδος, αναφυσβήτητα. Πολύ, πρέπει να το επενθυμίσουμε αυτό, να το υπογραμμίσουμε. Αλλά έχουμε κάποιους χώρους όπως ο μηχανισμός ελέγχου, όπως ελέγχθη προηγουμένως. Οι μηχανισμοί ελέγχου και το πεδίο εφαρμογής αυτοί οι δύο χώροι είναι αλληλένδετοι. Όταν υπάρχει διασαφήνιση ε, ε, ενός χώρου υπάρχουν κάποιες αβεβαιότητες έχουμε τα θέματα εθνικών αρχών που ανησυχούν σε σχέση με κάποια θέματα ε, ανταγωνισμών και αυτά θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε, να προβληματιστούμε ούτως ώστε όπως είπε η Ισπανίδα συνάδελφος που μας επενθύμησε ότι δεν θα πρέπει να, γίνει, να δημιουργηθεί ένα χάσμα ανάμεσα στο, στην αρμόδια αρχή και στο πολίτη για να μπορέσει να προστατευτεί ο πολιτής. Είναι σαφέστατα, θα πρέπει να υπάρχει μια γυτνίαση ανάμεσα, μια προσέγγιση ανάμεσα στον ε, πολίτη και στην ενίσχυση των ε, εθνικών αρχών ελέγχου στα πλαίσια φυσικά μιας ε, συνεργασίας που μου φαίνεται ότι είναι απαραίτητη στα πλαίσια αυτού του νέου δικαιώματος. Και να κλείσω λέγοντας ότι θα ήταν σημαντικό να υπενθυμίσω δηλαδή ότι από τη μια έχουμε την ε, αύξηση υπευθυνότητα στηριγμένη στην ε, εμπιστοσύνη αλλά που σήμερα απαιτεί διαφάνεια που δεν υπάρχει σήμερα στο κείμενο επίσης μια, ε, να γίνει ε, ένα σαφές το κείμενο, ε, το δίκαιο θα πρέπει να είναι δηλαδή ξεκάθαρο, κατανοητό από όλους και φυσικά χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο. Όσο πιο απλός είναι ο νόμος, τόσο καλύτερα εφαρμόζεται από όλους. Και να κλείσω τώρα υπενθυμίζοντας ότι σε αυτό το κείμενο τίθεται το θέμα της αποτελεσματικότητας. Αν υπάρχει μια αρχή η οποία θα λέγαμε έχει πολιτικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία φυσικά με τις διάφορες εθνικές αρχές, θα πρέπει ο στόχος μας να είναι, η αποτελεσματικότητα υπέρ του Ευρωπαίου πολίτη. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε στη θέση μας τεχνικά μέσα, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε ένα κείμενο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί, να είναι αποτελεσματικό τόσο σε, εθνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο γενικότερα, αλλά και στο εθνικό. Ευχαριστώ. Ήταν ε, πολλές οι ερωτήσεις, είπε στον κύριο Χόρνουμ. Οπότε έχετε και πάλι το λόγο και την ευκαιρία να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε δύο-τρεις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, εν συντομία, να πω ότι θα συμφωνήσω με τα επιχειρήματα του κυρίου Ράιχενμπαχ, ιδίω για τις ε, κοινότητες, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να συμπεριληφθούν αυτά, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει σε ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο του 21ου αιώνα και βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μέρο και του 21ου αιώνα και ε, τη κοινότητα. Οπότε εννοείται ότι θα επεξεργάζεται τα δεδομένα. Τώρα, για τι ερωτήσει που προσωπικά απευθύνθηκαν σε μένα. Πρώτον, νομίζω Κάποια ζητήματα ξεπέρασαν τα όρια του πεδίου της συζήτησή μας. Αλλά για το άρθρο 3, το πεδίο, δηλαδή την επικράτεια που καλύπτεται. Αυτό είναι μείζον ζήτημα. Πολύ σωστά εντοπίστηκε. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Νομίζω όμω ότι ω μείζον ζήτημα μπορεί να πετύσει και δύο, όχι μία, δύο γύρω συζήτηση, όχι μόνο έναν. Το πρόβλημα με το άρθρο 3 είναι για τον ελεγκτή, εν μέρη, μάλλον το πρόβλημα είναι αν ο ελεγκτή είναι στην επικράτεια τη Ένωση ή όχι. Η, η κατοικία των ατόμων για τα οποία συγκεντρώνονται τα δεδομένα. Εάν αποκλείσουμε κάποιε περιπτώσει, ίσω να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, αλλά θα πρέπει να προσδιοριστεί τι εννοούμε με την κατοικία, τι εννοούμε κάτοικο. Αυτό αυτό ούτω ή άλλω μέχρι τώρα ήταν κάτι που επιλειόταν σε επίπεδο κράτου μέλου. Ένα άλλο προβληματικό σημείο είναι τι σημαίνει προσφορά καλών υπηρεσιών σε άτομο για το οποίο συλλέγονται δεδομένα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αν ελεγκτή είναι εκτό Ένωση, στι ΗΠΑ λόγω χάρη, μπορεί να προσφέρει υπηρεσίε εντό Ένωση. Τι θα πει όμω προσφορά υπηρεσία προ κάποιον που βρίσκεται στην Ένωση αρκεί να υπάρχει ένας ιστότοπος ας πούμε όπου μπορεί καθένας να αγοράσει υπηρεσίες ε, από πουδήποτε αφορά τη γλώσσα αν θα χρησιμοποιούνται γλώσσες των κρατών μελών που κατανοούν οι πολίτες τους εδώ υπάρχει και το θέμα της ε, παρακολούθησης της συμπεριφοράς, διότι ο κανονισμός διέπει τους ελεγκτές οι οποίοι παρακολουθούν τη συμπεριφορά όσων κατοικούν εντός ένωσης λίγο πολύ. Δεν είμαι βέβαιος όμως τι ακριβώς μπορεί να εννοεί αυτό. Ε, δεύτερη ερώτηση. Για τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και για εταιρείες εντός και εκτός Ένωσης. Ναι, ναι. Θα συμβεί αυτό που λέτε. Διότι αν υπάρχει ένας αυστηρός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων εντός Ένωσης, βεβαίως ε, θα επηρεάζει τον ανταγωνισμό αν τα πράγματα εκτός είναι πιο χαλαρά. είναι κάτι που ούτω ή άλλω θα συμβεί. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι μείζον πρόβλημα και ποιε είναι οι εναλλακτικέ τώρα. Αυτό θα πρέπει να το μελετήσουμε. Τελευταία ερώτηση για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών επιβολή, και αν θα είναι όντω αποτελεσματική. Οι διατάξει για τι εθνικέ αρχέ προστασία των δεδομένων πραγματικά είναι βήμα πρόοδου. Οι αρχέ διευκρινίζονται με αρκετέ λεπτομέρειε προ την στιγμή και οι αρμοδιότητέ του τέλο πάντων είναι αρκετά συγκεκριμένε, αλλά ω προ το μηχανισμό συνεκτικότητα όχι. Όχι, διότι το βρίσκω επαχθέ ω μέτρο, χρονοβόρο και ήδη έχω σχολιάσει τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω. Θεωρώ πρέπει να βελτιωθεί το άρθρο 29. Η λεγόμενη αρχή για την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων, η οποία θα αποφασίζει για την ομιμότητα των περισσότερων υποθέσεων και μετά θα, θα επιλαμβάνεται το ΔΕΚ. Τώρα, η επιβολή πρέπει να στηρίζεται και σε κάποιες κυρώσεις. Οι διαδικασίες επιβολής όμως θα εξαρτηθούν και από τους πόρους που θα με τους οποίους θα προκοδοτηθούν οι Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων. Αυτό είναι κάτι που θα αποφασίζεται σε επίπεδο κάτω μέλους. Οπότε, ολοκληρώνοντας, να επισημάνω ένα ακόμη ζήτημα ο ρόλος των ιδιωτών κατά την διενέργεια ε, ε, ελέγχου, κατά τη λειτουργία των μηχανισμών. Για τους ιδιώτες, τι εννοούμε τώρα όμως με ιδιώτες, ακριβώς αυτούς για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα, τους πολίτες, τα δικαιώματά τους, τα, από τα πραγματικά τους δικαιώματα και τη διαφάνεια. Αλλά κατά τα άλλα, ιδιώτες και ο ρόλος των ιδιωτών μπορεί να σημαίνει και πάλι τη διασφάλιση διαφάνειας. Και ένα δεύτερο σημείο το οποίο έθιξε ο κύριος Ράιχενμπαχ. Οι ιδιώτες μπορεί να είναι και ανταγωνιστές. Μπορεί να αξιοποιούνται οι ανταγωνιστές μάλιστα εφόσον δέχονται τους ε, κανόνες προστασίας δεδομένων και θα μπορούσε και στον τομέα του δικαίου ανταγωνισμού να καλύπτονται ακριβώ και οι κανόνε προστασία δεδομένων, ώστε να καλύπτονται τα ίδια τα δικαιώματα των ανταγωνιστών. Θα μπορούσε δηλαδή να ασκηθεί και προσφυγή κατά κάποιου που παραβιάζει τα προστασία των ε, δεδομένων σε περίπτωση που υπάρχει ανταγωνισμός εμπορικός στη μέση. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γκονιέ να σας πω ότι ακόμη μπορείτε να ζητήσετε το λόγο. Έχουμε χρόνο. Έχουμε λίγο χρόνο προς το τέλος. Παρακαλώ, κύριε Γκονιέ. Ευχαριστώ. Ειλικρινά, ευχαριστώ τους βουλευτές. Είναι μοναδική ευκαιρία για να έχουμε ένα τέτοιο διάλογο. Με τιμά αυτό και είναι σημαντικό να δούμε τις, γνωμοδο... τις απόψεις των μεν και των δε, από την Ισπανία, από την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχουν όμως δύο σημεία πάνω στα οποία θα ήθελα να επανέλθω. Θα, ήθελα να έλθω σε ένα σημείο το οποίο είναι θεμελιώδος. Αυτό που έθιξε η βουλευτή από την Ισπανία. για το θέμα τη πραγματικότητα σε σχέση με την αρμόδια περιοχή που θα ε, αποφανθεί σε σχέση με τα δεδομένα και το θέμα της σύγκλησης ανάμεσα στην πραγματικότητα που έχουμε τώρα και το νέο κείμενο. Θα υπάρχει ένα θέμα που είναι το πιο βασικό. Εσείς είναι θυματικό αυτό που λέτε, αλλά και εσείς είσαστε που θα δώσετε μια απάντηση πώς θα μπορεί να συνδέσει κανείς να είναι σίγουρος δηλαδή ότι το νέο κείμενο που είναι ένας κανονισμός που έχει όλη αυτή την ισχύ. Πώς λοιπόν αυτός ο κανονισμός δεν θα βρίσκεται σε αντιπαράθεση σε σχέση που έχουν να κάνουν με την ε, ε, ιδιωτική ζωή. Εγώ δεν έχω απάντηση πάνω σε αυτό. Και, δεύτερον, και έχετε δίκιο, πώς θα γίνει ο πολίτης στην Ισπανία, Γερμανία, όπου αλλού στην Ευρώπη, να μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμά του. Πώς μπορεί να περάσει στην πράξη αυτό και από την άλλη πώς θα γίνει οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ε, έχουν όφελος από μια απλή διαδικασία. Θα πρέπει ε, να έχουμε ένα σωστό κείμενο, η εφαρμογή του δεν θα είναι εύκολη και, και ένας πολίτης δεν τον νοιάζει το θέμα της αναρμόνισης. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχει μια άμεση εφαρμογή ανεκειμένου και στο θέμα του μια άμεση απάντηση. Οι ερωτήσεις σας είναι σημαντικές. Σε αυτό όμως το στάδιο είναι ο νομοθέτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή που θα δώσει μια απάντηση. Είναι κάτι πάνω στο οποίο σίγουρα θα πρέπει να προβληματιστούμε. Θα υπάρξει διάλογο σίγουρα τις επόμενες μέρες. Το άλλο θέμα τώρα. Για την διαφάνεια. Η κυρία Σίπολα αναφέρθηκε ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να διασαφηνίσω αυτά που είπα. Πρέπει να γίνει σεβαστός ο νόμος. Τελεία Παύλα. Αυτού του λεχθέντος όμως είναι επίσης σωστό αυτοί οι οποίοι έχουν διάφορες δράσεις κοίταξα να σε γενικές γραμμές ο κύριος από τη Γερμανία αναφέρθηκε στο θέμα των κυρώσεων Χαίρομαι που υπάρχουν δυνατές μεγάλες κυρώσεις. Αναφέρονται θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτοί που δραστηριοποιούνται στον χώρο πρέπει να σέβονται το νόμο και αν δεν γίνεται αυτό να δεχθούν κυρώσεις. Και αυτές να ε, οι κυρώσει θα πρέπει να έχουν μια διαβάθμιση, διότι όλα δεν μπορούν να κυρωθούν με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, για την αποζημίωση. Εδώ θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα σε σχέση με το άρθρο 39 του υπάρχοντος κανονισμού, διότι πριν από λίγο να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα τα άρθρα 38-39 με τον τρόπο συμπεριφορά είναι κάτι για το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα το αναπτύξουν επιχειρήσει. Αυτό που χρειάζεται σήμερα, και εδώ έχουμε να κάνουμε τα κίνητρα, δηλαδή μια επιχείρηση θα πρέπει να έχει ένα κίνητρο. Σήμερα δεν το έχει. Διότι ο, ο μηχανισμός που που λέμε πηγαίνει αργά-αργά, ίσως αργότερα σε μερικά χρόνια να βελτιωθεί. Αυτό το θέμα της συμπεριφοράς θα πρέπει να διασαφηνθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον όμως σε ευρωπαϊκό, διότι ξέρω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Έχουμε ένα προϊόν Φερρυπίν το οποίο αναπτύσσεται σε, μια, σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας Ε, το οποίο ε, έχει ένα αλφα κόστος. Ένα προϊόν το οποίο δεν αναγνωρίζεται καν σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Σκεφτείτε τώρα τι θα γίνει όταν έχουμε κάτι σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα. Διότι όταν κάνει μια επιχείρηση μια προσπάθεια θα πρέπει να έχει και κίνητρα σε σχέση με τη ε, διαφάνεια αυτό που θα ήταν καλό είναι να έχουμε και κίνητρα για την ανάπτυξη προϊόντων τα οποία έχουν να κάνουν μια προσέγγιση διαφανή και θα μπορούσα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Microsoft για όλα τα προϊόντα δημιουργεί ένα κέντρο. Ένα κέντρο στο οποίο υπάρχει εμπιστοσύνη. Το λεγόμενο Trust Center. Άλλες εταιρείες δεν ξέρω που το κάνουν αλλά προτείνω και άλλες εταιρείε να το κάνουν. Για να, δείχνει, να εξηγούν πού ακριβώς καταλήγουν τα δεδομένα. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αξιολογούνται ε, όταν, όταν και πώς το κάνουν αυτό, διότι δεν καταλήγουν πουθενά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια αναγνώριση για αυτήν εδώ την προσέγγιση και θα περιοριστώ σε αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ροδρίκε, νομίζω υπάρχουν ερωτήσει ε, που αφορούσαν εσά ε, απευθεία. Σας πρέπει να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στη μονοθυριδική προσέγγιση και τις ανησυχίες ότι ο καταναλωτής, ο πολίτης δεν θα έχει ευχερή πρόσβαση και δυνατότητα αποκατάσταση των προσωπικών του δεδομένων ή ε, προστασία από την αρμόδια αρχή. Η μονοθεριδική προσέγγιση νομίζω είναι μια καλή λύση. Αλλά Πρέπει να είναι απόλυτα σαφή η κατάσταση. Και το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρωί ότι την ισχύει ιδιαίτερο στο γεγονό ότι και αυτή η μονοθυρητική προσέγγιση ενδεχομένω να μην δίνει την απάντηση, δηλαδή να μην εκπροσωπείται ο πολίτης από την αρχή την αρμόδια για την δεδομένων της χώρας κατοικία ή διαμονή. Άρα Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, θα πρέπει δηλαδή να είναι σε θέση να προσφεύγει στην αρχή τη χώρα διαμονή του ο πολίτη. Ένα, αυτό πρέπει να είναι απόλυτα σαφέ δικαίωμα. Και δεύτερον, έτσι ώστε οι αρχές προστασίας δεδομένων να είναι σε θέση να χειριστούν, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, θα πρέπει να είναι σε εντατική συνεργασία μεταξύ τους. Μπορεί να μην υπάρχει αυτή η πρόταση, αλλά πιστεύω ότι η δικτύωση που ήδη υφίσταται, πρέπει να αξιοποιηθεί και πρέπει να διδαχθούμε από την εμπειρία ε, που μας προσφέρουν τα εφιστάμενα δίκτυα αρχών προστασίας δεδομένων που έχουν θεσπιστεί εδώ και μερικά χρόνια. Το δικαίωμα για το καταναλωτή, του υποκειμένου θα λέγαμε του δικαιώματος αυτού, να προσφύγει σε μια ε, αρχή, στην κατάλληλη αρχή, έχει τεράστια και κρίσιμη σημασία. Επίσης, άλλη ερώτηση που αφορά την προστασία δεδομένων, προσωπικών δεδομένων παιδιών, ανηλίκων. Εδώ υπάρχει μια πρόταση. για την οποία επισημάνθηκε από κάποιον από το ακροατήριο ότι μπορεί να γεννά πολλές δυσκολίες. Όντως, θα πρέπει το profiling των παιδιών να απαγορεύεται τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών να προστατεύονται Η απαγόρευση ωστόσο στην πρόταση όταν έχουμε να κάνουμε με την εφαρμογή, όταν έρθει η ώρα της εφαρμογής μπορεί να οδηγήσει δυσκολίες. Γιατί, Γιατί το έτος της ενηλικίας διαφέρει από, έτος, από κράτος σε κράτος. Άρα τι σημαίνει παιδί. Και δεύτερον, μπορεί να οδηγήσει στην ε, επεξεργασία περισσότερων ακόμη δεδομένων εισαγωγή αυτή τη διάταξη. Άρα χρειάζεται βεβαίω ναι, συνένεση ως προς την, και γενικά αποχώρηση ω προ την επεξεργασία δεδομένων ανηλίκων, αλλά θα πρέπει και να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε κατάλληλα τεχνικά μέσα ώστε αυτή η διάταξη να μην οδηγήσει ακόμη περισσότερα δεδομένα που θα διατίθενται για επεξεργασία, δεδομένα παιδιών. Τρίτον, το δικαίωμα στη λύθη και συμβατότητα ή ανάγκη για εξέβρεση ισορροπίας σε ορισμένες περιπτώσεις ως προς την ελευθερία έκφρασης. Δεν θα είναι σαφές για μένα αυτό που ενώσατε με την ερώτηση σας. Δεν ξέρω αν ε, θέλετε να το επαναλάβετε ή αν αναφερόσασταν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Η προσέγγιση προσωπικών δεδομένων πάντως έχει προφανώς όρια που μερικές φορές έχουν φτάσει μέχρι τα δικαστήρια για να προσδιοριστούν και θα πρέπει να αναζητηθεί αυτή η ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ιδιαίτερα δε εδώ με, την, ε, με το δικαίωμα στη λύθη. Τώρα, εάν έχετε κάποια επιπλέον... Ο κύριος Σκέλη νομίζω το έχει ζητήσει αυτό, το έχει ρωτήσει αυτό. Ο κύριος Σκέλη αν θέλετε να επαναλάβετε την ερώτηση. Θέλετε να λάβετε το λόγο κύριε Κέλλη. Όχι. Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέει ο πρόεδρος και ο κύριος Ντέιβις για να απαντήσει σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ στόμα. Και την τελευταία ερώτηση που ακούστηκε φθηνόμενη σε μένα της απεριόριστης έκτασης της συλλογή δεδομένων, απεριόριστης έκτασης κατά ε, την υποβολή ετοιμάτων για χορήγηση προσωπικών δεδομένων από τον πολίτη. Εγώ θα σας επισημάνω ένα στοιχείο που έχω, ότι μέχρι τα 16 του χρόνια ένας ε, πολίτης έχει ήδη διαθέσει το μεγαλύτερο ποσοστό των προσωπικών του δεδομένων. Μέχρι τα, 20, μέχρι τα 18 το κράτος έχει συλλέξει ό,τι επέμενε και ως εκ τούτου μέχρι τα 21 του ένας πολίτης το πολύ πολύ να έχει διαφυλάξει κάποιες προσωπικές στιγμές που μπορεί ένας από τους ε, ερωτικούς του συντρόφους να έχει φυλάξει και να μην έχει δημοσιοποιήσει. Αυτό είναι ότι μένει από το προσωπικό ιδιωτικό βίο δηλαδή. Άρα, έχουμε αιτήματα μιλάτε για μονοθυριδικές ε, λύσεις. Άλλωστε θα πρέπει να βρούμε σαν λύση την μονοθυριδική ταυτότητα, την ε, μονοθυριδική, ε, το μονοθυριδικό διάβλο ή την επικοινωνία, τη δικτύωση. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίσαμε στον εμένα Βασίλειο ιδιαίτερα με την μεγάλη συζήτηση και το δημόσιο διάλογο για την ε, ταυτότητα, για το δελτίο ταυτότητας που, που αποφασίστηκε να εκδοθεί εν τέλει. Αυτό, είναι μια καταστρο... Αυτό ε, λοιπόν μπορεί να οδηγήσει σε μια καταστροφή ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη εάν προχωρήσει με τον τρόπο με τον οποίο έχει προταθεί. Χρειάζεται λοιπόν να αναλογιστούμε και πάλι τον κανονισμό με καινοτόμες λύσεις όπως η Μάιντεξ επί παραδείγματος του Ηνωμένο Βασίλειο που προσπαθεί να με τα φορτώσει πολλές από τις προνομίες και τις εξουσίες το είναι ίδιο το, τον ιδιώτη, το άτομο δηλαδή. Αυτή είναι μια από τις καινοτομίες που ε, υπάρχουν στην Ευρώπη και στο γενικότερο κόσμο ε, αλλά που αγνοούνται ή παραγνωρίζονται καλύτερα και προτιμούνται στη θέση τους μεγάλες ε, λύσεις, ογκώδεις λύσεις, βαριές λύσεις που έχουν να κάνουν με τον επιχειρηματικό κόσμο. σε ένα ερώτημα το οποίο μπορώ να παραφράσω εξή πώ μπορεί να χωνέψει η Ευρώπη τα όσα πράττονται εδώ, τα όσα πράτετε εσείς. Εγώ δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μια απαξία στην ιδέα της, ε, προσωπικής, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τις εθνικές αρχές. Δεν εννοώ ότι έχουν απαξιωθεί εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων. Αλλά όπως και να έχει υπάρχει μια απογοήτευση από πλευράς του κοινού. Αυτό όμως δεν ε, σχετίζεται απαραίτητα με τη συμπεριφορά της ε, υπηρεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του, ε, της κυβερνήσεως, με την νομοθεσία, με τη γενικότερα και περιραίουσα ατμόσφαιρα περί μεγάλου αδελφού. Γενικά οι, προσωπι... οι ε, υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων χαίρουν ιδιαίτερη εκτίμηση από τους πολίτες των χωρών τους. Ίσως όμως, ίσως όμως θα ήταν ένα θέμα αυτό το οποίο θα μπορούσε να προβληθεί και σε ε, περιπτώσεις φερρυπίν εκλογικών αναμετρήσεων. Θα μπορούσε ένας υποψήφιος να προβάλλει την ιδέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ως μια σημαντική αξία που προάγει. Ωστόσο, μένουν άλλα ερωτήματα από τα οποία δεν απαντά αυτό ο κανονισμό. Το πώ αντιμετωπίζονται, παραδείγματι, οι υπεράκτιε εταιρείε διαχείριση δεδομένων ή διάφορε άλλε εταιρείε που χωρί να θέλω να δώσω ονόματα, ε, μαθαίνουμε από τα νέα, από τι ειδήσει, από τι τηλεοράσει ε, και τα γνωρίζει όλο ο κόσμο βεβαίω, ότι παραβιάζουν ε, κατάφορα ορισμένε διατάξει περί προστασία ε, προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη και κυρίω εδώ αναφέρομαι βέβαια σε αμερικανικέ εταιρείε που αδράχνουν τι ε, αδράτουν τις πληροφορίες και έτσι εκμεταλλεύονται. Άρα λοιπόν χρειάζεται περισσότερη λεπτομέρεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ε, πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε μια ουσιαστική ρύθμιση ε, και όχι μια ρύθμιση στο πόδι, μια γενικόλογη ρύθμιση. Για να μπορέσουμε να κερδίσουμε, αν θέλετε να κερδίσετε εσείς τον πολίτη, είναι σημαντικά τα ζητήματα αυτά. Και μια τελευταία παρατήρηση, εδώ δεν μιλάμε για ένα κανονισμό περί εκδόσεως ε, κατηγορουμένων ε, ποινικών εγκληματιών. Εάν όμως ήταν αυτός ο, ένας κανονισμός περί εκδόσεως, είμαι βέβαιος ότι θα συζητούσαμε και θέματα αμοιβαιότητας και θέματα ε, εκ πρώτης όψης αξιολόγησης των συνθήκων και θέματα προληπτικής προστασίας και όλα αυτά. Επομένως είναι θέμα το οποίο αφορά στην ουσία της τη ζωή του πολίτη και αυτό που δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε, και στο συγγνώμη αν σας κάνω κήρυγμα από αυτή τη θέση, είναι ότι δεν έχουμε κερδίσει τον πολίτη. Αυτό πρέπει να καταφέρουμε λοιπόν, να πείσουμε το μέσο πολίτη ότι αυτό που κάνουμε είναι για το καλό του. Ευχαριστώ πολύ. Μας έχουν μείνει μερικά λεπτά μόνο για τη Βαρόνι Λάτφορτ από τους φιλελεύθερους δημοκράτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα σχόλια μόνο Να ευχαριστήσω τον κύριο Ντέιβις. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβει μέρος και στην προεκλογική εκστρατεία για το 2014. Μας έδωσε πολλές καλές ιδέες για να ξέρουμε τι να ισχυστούμε. Για την κατάρτιση προφίλ τώρα, ήδη πριν από 3,5 χρόνια, στο τέλος της προηγούμενης θητείας, το συζητήσαμε με μια έκθεση πρωτοβουλίας η οποία θα αποτελούσε μέρος ενός προγραμματιζόμενου νομοθετήματος, αλλά δικαίως το έθεσε κ. Γκόνιε. Υπάρχει εδώ μια αιμονή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι μπορεί να αρνηθεί κανείς την κατάρτιση προφίλ μόνο αν υπάρχουν νομικές συνέπειες και όχι στην κατάρτιση προφίλ αυτή καθεαυτή. Ελπίζω ότι είναι κάτι που θα αντιμετωπιστεί. κατά την όλη επεξεργασία του κανονισμού. Υπάρχουν πολλέ περιπτώσει που μπορεί να προκύψουν. Δεν λέω ότι όλε οι περιπτώσει κατάρτιση προφίλ πρέπει να απορρίπτονται, αλλά η κατάρτιση αυτή καθεαυτή θα πρέπει να ρυθμιστεί. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις που μπορεί να προκύψει βλάβη, δηλαδή, να παραβιάζεται ο ιδιωτικό βίο, ακόμη και να μην, χωρίς να υπάρχουν ε, άμεσες άμεσε νομικέ συνέπειε η καθολου νομικέ συνέπειε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ε, κάθε φορά που κάποιο πρόβλημα προκύπτει επιμένει. Πρέπει να απορρίπτεται η κατάρτιση προφίλ μόνο αν προκύπτουν συγκεκριμένες νομικές συνέπειες. Ούτε οι εθνικές κυβερνήσεις ε, εμποδίζονται στο να κάνουν, ε, να, να καταρτίζουν προφίλ, αλλά σε αντιδιαστολή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον το αναγνωρίζουν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για αυτή την τελευταία παρέμβαση. Δεν ξέρω αν θέλουν ε, τα μέλη του πάνελ να κάνουν κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Απλώς θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι όσο θέλετε. Κύριε Γκονιέ, ένα λεπτό. Να περάσω στα γαλλικά, αν και αυθορμήτως απαντάω αγγλικά. Ευχαριστώ όλους που πήραν το λόγο για την ευκαιρία που μας έδωσαν να παρουσιάσουμε και εμείς τις δικές μας απόψεις. Εκπροσωπήθηκαν ε, πολλές χώρες και αυτό είναι θετικό. Αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας συγκεκριμένος ρυθμός. Ένας ρυθμός και η στιγμή αυτή, η συγκυρία που ζούμε είναι καταπληκτική. Έχετε το ρόλο σας ως βουλευτές και ευρωβουλευτές, θα αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία τα επόμενα χρόνια, νομοθετικό ρόλο μάλλον, αλλά να μην ξεχνάμε και το προηγούμενο ζήτημα, το παράδοξο παιδιωτικού βίου. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης ξέρει ότι είναι ιδιωτικός βίος. Αυτό να μην ξεχνάμε. Τα δεδομένα που περνάνε σε όλα τα κανάλια, στο διαδίκτυο καθημερινά. Τα γνωρίζει ο Ευρωπαίος πολίτης ότι αποτελούν μέρος του ιδιωτικού του βίου. Ο ιδιωτικός βίος, ο ιδιωτικό βίο έχει κάποια αξία. Τα δεδομένα έχουν κάποια αξία. Γι' αυτό θα πρέπει να ενημερώσουμε του Ευρωπαίου πολίτε. Αυτό είναι πραγματική πρόκληση. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρο. Ευχαριστώ για τι τελευταίε κυρία ευχαριστώ πολύ το κοινό, τους διοργανωτές. Συμφωνώ με τον παρακαθήμενο ότι είναι πολύ σημαντικό η πρόταση του κανονισμού έχει κέρια σημασία ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις ε, με κάποιο τρόπο παρακολουθούνται και υπάρχουν ε, διασφαλιστικές δικλείδες. Ίσως δεν είχαμε αντιληφθεί πόσο γρήγορα προχωράει αυτή η εξέλιξη τεχνολογική και πόσο βραδία είναι η πορεία της ε, νομοθεσίας. Πρέπει λοιπόν και βέβαια με φρόνηση και σύνεση να σπεύσουμε βραδέως θα έλεγα ή ταχαίως καλύτερα στην, στο νέο αυτό νομοθέτημα, το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες για τους καταναλωτές, τα υποκείμενα δηλαδή δικαίου, δικαιώματος, εισάγονται νέα δικαιώματα για τη διαφάνεια, νέα συνθήκες για πρόσβαση, νέα δικαιώματα για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων σε περίπτωση παραβίασης και αναφέρθηκε και το πρωί βεβαίω ότι η πρόταση εν όλο είναι πολύ θετική, ωστόσο κάποια ζητήματα πρέπει να προσδιοριστούν, να διευκρινιστούν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει βεβαιότητα ασφάλεια δικαίου ουσιαστικά για τον επιχειρηματή αλλά και για τον καταναλωτή και ε, επισημαίνω ότι υποστηρίζουμε μεγάλο, σε κάποιο βαθμό τα σχόλια των ε, άλλων ομιλητών ως προς τον ε, τεράστιο ρυθμό των ε, δεδομένων που διαβιβάζονται ή που τυχάνουν επεξεργασίες και η Επιτροπή θα ήθελα να σας πω με τις εκτελεστικές της εξουσίες προσπαθεί να δώσει λύσεις. Κάποιες όμως από τις προβλεπόμενες πράξεις ε, ίσως είναι ίσως ξεπερνούν αυτές τις εξουσίες θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ποια από τα δεδομένα αυτά εντάσσονται στα θεμελιώδη δικαιώματα και σε ποιο βαθμό μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, Πρόεδρε, ο κύριος Δέβης, πολύ σύντομα και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω την πρωτοβουλία πρέπει να αξιολογηθεί ως ευκαιρία περισσότερο, χρειάζεται περισσότερη καινοτόμα προσέγγιση Πάντω θα ήθελα να πω με μια παράκληση, με όλη τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα και τι ευκαιρίε που υπάρχουν, αυτή η ιδέα της ασφάλειας, της συνέπειας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας πρέπει να καταστεί ιερό σύνθημα για, την, ε, για τον νομοθέτη, για την ε, καταδεξιοδότηση νομοθετική πράξη κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης ε, θα συνεχιστεί η έρευνα που κάνουμε με τους εμπλεκόμενους, τους stakeholders. Γι' αυτό όποιος ενδιαφέρεται παρακαλώ να έρθει σε επαφή μαζί μου το τέλος της σα. Θα ήθελα, επί τη ευκαιρία, μια και ο πρόεδρος έχει θέματα ε, τεχνολογίας, ε, μάλλον νομικών, νομικών θεμάτων ή δικαίου των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά με το μέλλον της προστασίας στο ίντερνετ για το μέλλον. Χρειάζεται ασφαλώς ε, η προστασία, χρειάζεται η εποπτεία, οι developers, αυτοί που θα αναπτύσσουν δηλαδή την ε, τεχνολογία, αλλά και αυτοί που θα την επαληθεύουν. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και προστασία του ιδιωτικού βίου σχεδιασμένη κατά περίπτωση δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά, λέει ο Πρόεδρος, και την κυρία Μαριέτα Καραμαντλή, η οποία δυστυχώς χρειάστηκε να αποχωρήσει νωρίτερα, το είδατε ασφαλώ. Πιστεύω ότι έτσι έχουν ε, διευκρινιστεί κάποια σημεία της συζήτησης. Θα δούμε και κάποια άλλα αργότερα σήμερα και αύριο. Σας ε, υπενθυμίζω μόνο ότι τρεις ακριβώς ε, το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με την ομιλία, εναρκτήρια ομιλία της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίας Βιβιάν ε, Ρέντινγκ. Και όποιος εξημών θέλει να δει λίγο περισσότερο τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, έχουμε τρία έγγραφα εργασίας που παρουσιάζονται σήμερα. Τα βλέπετε εδώ στα δεξιά της έδρας, βγαίνοντα δηλαδή από την πόρτα. Έχουν να κάνουν με τον κανονισμό και με την οδηγία τα έγγραφα εργασίας και μετά την κήρυξη του πέρατος αυτής της ε, ε, συνεδρίας έχουμε μία μικρή δεξίωση για τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και για τους ομιλητές της έδρας. Μία δεξίωση εδώ στην ε, είσοδο. Σας ευχαριστώ όλους.